Yeah, yeah, Good um, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινήσουμε στην ώρα μας ε, γιατί έχουμε έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο σήμερα μαζί μας σε μία από τις τελευταίες ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Ας ξεκινήσουμε με κάποια τυπικά ζητήματα. Έγκριση της ημέρησιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να εγκρίνουμε χωρίς τροποποίηση της ημέρησιας διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Σε 15 γλώσσες έχουμε διερμηνία και η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά τώρα της συνεδρίασης της 12 η Ιανουαρίου είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό επιγραμμικό φάκελο. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις σχόλια θεωρώ ότι εγκρίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Μπιενκόφσκα, την επίτροπό μας μπορώ να πω. Έχουμε δει πολλούς επιτρόπους και πρώην επιτρόπους, εσείς είστε η δική μας πάντως επίτροπος, στα πλαίσια της εξαστικής αυτής επιτροπής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό συνοψίζοντας όλες αυτές τις ακροάσεις που διοργανώσαμε να σα ακούσουμε για ακόμα μία φορά, για μία ανταλλαγή απόψεων αυτή τη φορά, όχι για λόγους ακρόαση. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που θέλουμε να καλύψουμε, όχι μόνο για το παρελθόν και την υποεξέταση έκθεση, την οποία θα καλύψουμε εκτενέστρα και μετά την παρέμβασή σας κύριε Επίτροπε, αλλά να δούμε και λίγο όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Να δούμε δηλαδή πώς θα καλύψουμε τον τρίτο καονισμό της Επιτροπής σχετικά με τις εκπομπές της συνθήκης πραγματικής οδήγησης, τι θα γίνει με την πρόταση για τις αρχές έγκρισης τύπου, μια πρόταση η οποία θα εγκριθεί αν δεν κάνω λάθος να ψηφιστεί σήμερα το πρωί. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσοι ήρθαν από την ΙΜΚΟ στην Επιτροπή αυτή και από τη δική σας τη Γενική Διεύθυνση, γιατί πραγματικά συνέβαλαν πάρα πολύ στο να καταφέρουμε εμείς να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πορίσματα, συμπεράσματα και συστάσεις, ιδίως όσον αφορά το σύστημα έγκρισης τύπου. Εμείς θέλουμε να βαθμίσουμε σαστικά τις αρχικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε τις δύο αυτές εκθέσεις στην Ολομέλεια και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσουμε να ασκούμε πίεση στο Συμβούλιο. Λοιπόν, για να είμαι σαφής, δεν πρόκειται για ακρόαση, πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων. Δίνω το λόγο τώρα στην Επίτροπο την κυρία Μπιενκόφσκα για να κάνει κάποιες εισαγωγικές παρεμβάσεις και συνέχεια θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, τους συνεισηγητές μας και θα ακολουθήσει και τη δικασία Catch the Eye. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο το τι γίνεται τώρα. Να σας ευχαριστήσω για το έργο αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής γιατί δεν υπερβάλλω αν πω ότι η δουλειά σας με βοήθησε να προχωρήσω σε πολύ σημαντική νομοθεσία και βεβαίως θα συνεχίσετε να με βοηθάτε και στο επόμενο βήμα. Διάβασα βέβαια το σχέδιο έκθεσης και τις συστάσεις και περιμένω να διαβάσω την τελική έκθεση. Τώρα έχει περάσει 1,5 χρόνος βέβαια μετά τις πρώτες αποκαλύψεις. Πολλή δουλειά έγινε για να καταλάβουμε τι συνέβη και γιατί και για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Παρά τις προσπάθειες αυτής της Επιτροπής και της Κομισιόν, ακόμα προσπαθούμε να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία από τις εθνικές έρευνες. Όταν μιλάμε με πολλούς εκπροσώπους του κλάδου, νομίζω και εσείς το έχετε ζήσει αυτό, και εγώ και εσείς, βλέπουμε πολλές φορές μια άρνηση. Δεν υπάρχει λοιπόν αλλαγή στάσης ε, ε, στον κλάδο, αλλά δυστυχώς ε, και στις αρχές των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη ακόμα αρνούνται να μας αποκαλύψουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στα πλαίσια των εθνικών ερευνών. Η γενική λοιπόν στάση δεν έχει αλλάξει και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι όπως ε, έχω επαναλάβει πολλές φορές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ούτε μπορούμε να βοηθήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία αν δεν έχουμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ελπίζω ότι η έκθεσή σας θα το αναγνωρίσει αυτό. Η Επιτροπή σας συμβάλλει με τρόπο πολύτιμο γιατί έτσι θα χυθεί φως στα όσα συνέβησαν και βεβαίως θα δει ο καθένας τις ευθύνες του. Ε, εμείς προσπαθήσαμε, ελπίζω να γίνει αυτό ε, κατανοητό ότι προσπαθήσαμε εμείς ως Κομισιόν να βοηθήσουμε στα πρώτα βήματα και να επιλύουμε προβλήματα. Η Επιτροπή συμπληρώνει τη δική μας τη δουλειά για να δούμε τι πήγε άσχημα και πώς θα διορθωθεί. Η έκθεσή σας αντιλαμβάνομαι ότι θα επικρίνει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προσωπικά και όλοι σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας Δύο πράγματα όμως πρέπει να πούμε. Ενώ όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα, ε, δεν θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα χωρίς ε, την βοήθεια του κλάδου και των ε, αρχών των κρατών μελών. Ε, και όπως σας είπα δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη ακόμα. Ελπίζω αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην τελική σας έκθεση. Και περνώ στην ουσία αυτό που θέλω να πω σήμερα. Πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον. Οι δράσεις μας πρέπει να κάνουν καλύτερα τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν σωστές αγορές, να έχουν εμπιστοσύνη στα αυτοκίνητα που αγοράζουν και οδηγούν και βέβαια να συμβάλλουν και στους περιβαλλοντικούς μας στόχους και τους στόχους μας για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα θα πρέπει ο κλάδος να παραμείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο αλλάζει ταχύτατα. Ξέρετε ότι εργάστηκα στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε τρεις τομείς. Καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας, καλύτερη εποπτεία της αγοράς, καλύτεροι κανόνες. Να τονίσω επίσης ότι το έργο της Επιτροπής σας ήταν κεντρικής σημασίας, το τονίζω αυτό, γιατί με βοήθησε να προχωρήσω και στους τρεις μου στόχους. Καταρχήν, εγώ αντιμετωπίζω πάρα πολύ δυναμικά το θέμα της επιβολής της νομοθεσίας και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας εδώ. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση, όπως ξέρετε, ε, κατά 7 κρατών μελών. Το Δεκέμβριο έγινε αυτό, διότι δεν εφάρμοσαν τους κανόνες έγκρισης τύπου των οχημάτων, ακόμα υπάρχουν ανεπαρκείς κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων στις χώρες αυτές, αλλά νομίζω ότι δεν τελειώσαμε τη δουλειά μας εδώ, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες παραβάσεις. Είμαστε ακόμα σε επαφή με άλλα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε τα δικά του συστήματα και αν χρειαστεί θα, θα γίνουν και άλλες διαδικασίες επί παραβάση, δεν μπορώ να σας πω πότε, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν παραβάσεις. Δεύτερον, όπως λέει πολύ σωστά το σχέδιο έκθεσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εποπτεία της αγοράς. Εμείς ε, δράσαμε σε δύο μέτωπα. Καταρχήν υποχρεώσαμε τα κράτη-μέλη να μας ενημερώνουν Εμά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι προσπάθειε που κάνουν για την εποπτεία τη αγορά και ε, ό,τι αφορά την επιβολή του νομοθετικού πλαισίου στην νομοθετική μα πρόταση για την έγκριση τύπου. Τέλος, ε, πρόκειται για πρακτικέ βελτιώσει βελτιώσεις επιτόπου. Δηλαδή να υπάρχει αποτελεσματική και ανεξάρτητη υποπτία της αγοράς. Τρίτον, χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες όχι μόνο για την υποπτία της αγοράς, αλλά συνολικά, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζει η εκθεσή σας. Έτσι λοιπόν έχω υποβάλει ε, σχέδιο κανονισμού για να βελτιώσουμε ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και κατανάλωση καυσίμων. Ε, έχουμε ολοκληρώσει μια νέα πολύ στεναρή ε, διαδικασία για να δούμε τις δοκιμές εν κινήσει. Η τέταρτη και τελευταία πράξη, θα ασχολείται με τις δοκιμές αυτοκινήτων εν χρήση. Ε, που ε, ε, χρησιμοποιούνται δηλαδή. Επίσης ανταποκρίθηκα στην πρόταση σχετικά με τις διατάξεις αναστολής. Θα πρέπει δηλαδή να ε, τηρούνται όλοι οι κανόνες. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι προτείναμε ένα πολύ πιο στεναρό σύστημα για την έγκριση τύπου. Τα κράτη-μέλη ήθελαν να ε, αποκλείσουν την αρμοδιότητα ε, απαγόρευσης ε, και κυρώσεων στους κατασκευαστές. Πριν από ένα χρόνο είχα κάνει μια πρόταση για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση να αντιμετωπίσουμε κακοδιοίκηση σε εθνικό επίπεδο και βέβαια σημαντικό θα είναι να αποκαταστήσουμε και την ε, εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης. Το έχω πει πολλές φορές, η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και η Επιτροπή σας και γενικά το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ζήτημα το βασικό είναι να συνεργαστούμε εν προκειμένου και αυτό είναι το κύριο αίτημά μου προς εσάς ε, κυρία Πρόεδρε ε, όπως ε, είπαμε, ελπίζω να οι συνάδελφοι στην Επιτροπή ΙΜΚΟ να ε, συνεργαστούν με το έργο της ειδικής σας της Επιτροπής, να υπάρξουν ε, ε, από κοινού προτάσεις και βασίζομαι σε εσά αλλά και στους συναδέλφους σας να αντισταθείτε σε οποιαδήποτε πρόταση αποδυνάμωσης της, της πρότασης της Επιτροπής πριν από ένα χρόνο. Βέβαια, ε, και οι διαδικασίες στο Συμβούλιο είναι ε, αργές. Θα ήθελα να κάνει περισσότερες προσπάθειες η Μαλτέζικη Προεδρία. Τους ζητήσαμε να επιταχύνουν τις διαδικασίες ε, στα πλαίσια της ε, συζήτησης και έγκρισης της έκθεσης για την, της πρότασης για την έγκριση τύπου. Είναι σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα και ουσιαστικά όμως. Τα επόμενα χρόνια θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, γι' αυτό αρχίσαμε και τη διαδικασία 2030. Είμαστε τώρα πιο κοντά ε, στις ε, ε, ε, νέες αλλαγές ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Θα μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε και τη ζωή των πολιτών, αλλά υπάρχει και μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αυτές οι αλλαγές θα επιφέρουν και πρακτικές αλλαγές, δηλαδή θα υπάρχει μεγαλύτερη περιπλοκότητα στα αυτοκίνητα, οπότε είναι σημαντική η κοινωνική αποδοχή, η εμπιστοσύνη. Αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εκπομπών, να εργαστούμε Εγώ ε, είμαι στο τέλος της ε, ομιλίας μου. Ε, θα σας το τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα αναδείξατε και αποκαλύψατε στο σχέδιο έκθεσης. Ε, ευχαριστώ πολύ και βασίζομαι σε σας και για το μέλλον, γιατί έχουμε καθυστερήσεις και θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θα δώσω το λόγο στους δύο Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κυρία Μπιενκόφσκα στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι ακρόαση, είναι ανταλλαγή απόψεων. Καλωσορίζω αυτά που είπατε αρχικά. Αναφέρατε πολλά πράγματα για την προστασία των καταναλωτών, ε, για μια δίκαιη συμφωνία περί μιλήσατε για τις παραβιάσεις στα κράτη-μέλη, είπατε ότι ενδεχομένως ε, κι άλλες αποκαλύψεις θα γίνουν σε σχέση με κακοδιοίκηση. Ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι δύσκολο ε, είναι ότι πολλές φορές συζητούμε για την έγκριση τύπου και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ε, ε, υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, συναλλαγών ύψους πολλών εκατομμυρίων στην Ευρώπη σε αντίθεση με την Αμερική δεν έχουμε ενιαία βάση για αποζημιώσεις. Στην Ευρώπη τα οχήματα και της Volkswagen μπορούν να ε, επισκευάζονται. Αν δεν υπάρχει ενιαία ε, ε, νομική βάση, πώς μπορούμε να ζητήσουμε ενιαία αποζημίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα πρέπει να, είναι, να υπάρχει ένα fair deal, αλλά χωρίς να υπάρχει απαραίτητη νομική βάση, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μπορούμε να πάρουμε κι άλλες όλες τις ερωτήσεις μαζί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι περίμενα να σχολιάσετε το σχέδιο έκθεσής μας. Ίσως μπορείτε να το κάνετε αργότερα όταν μας απαντήσετε. Πρέπει να το πω όμως ότι περίμενα κάτι να πείτε γι' αυτό, ένα είδος με ακούλπα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Συμφωνώ πολύ με ό,τι είπατε στα εναρκτήριά σα σχόλια. Είναι σαφέ όμως ότι πρέπει να εντοπιστούν σαφείς περιπτώσεις ε, ε, κακής διοίκησης και κακής διαχείρισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Ωστόσο, ας μην το δούμε σήμερα, έστω. Γιατί εξεπλάγει με τα σχόλιά σας σήμερα το πρωί. Είπατε και ο κλάδος και τα κράτη-μέλη δεν έχουν αλλάξει στάση. Και αυτό με άφησε άφωνο. Είναι από τις πιο καταπληκτικές δηλώσεις που έχω ακούσει σε αυτή την Επιτροπή. Ε, πραγματικά έχω μείνει άναυδος γιατί λέτε ότι ε, τα κράτη-μέλη δεν κατανοούν και συνεχίζουν να μην κατανοούν πόσο καταστροφικό είναι αυτό το σκάνδαλο το Dieselgate και πόσο θα είναι και στο μέλλον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Από την άλλη, μπορεί να μένω άναυδος, αλλά άναυδος δεν σημαίνει και έκπληκτος, γιατί βλέπω ότι παραμένει ε, η τακτική των κρατών μέλων. Δεν μοιράζονται τα στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που θα έπρεπε. Βλέπω ότι οι εθνικές αρχές δεν αναλαμβάνουν τη δράση που χρειάζεται. Και παρατηρώ ότι ο κλάδος, η αυτοκινητοβιομηχανία, συνεχίζει να αρνείται τις ευθύνες της. Και όχι μόνο η Volkswagen. Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Βλέπω και πολύ φοβούμαι ότι όλοι βλέπουμε τις τεράστιες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης εδώ. Εάν δούμε τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι ΗΠΑ εναντίον της Volkswagen, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Διαπιστώνουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε επέβαλαν τον νόμο, τον εφάρμοσαν και κατάφεραν να αποφύγουν ο κλάδος να εξαπατήσει στο μέλλον. Ε, κατάφεραν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, οι οποίοι ε, έγιναν αντικείμενο ε, κοροϊδίας και εξαπάτησης από αυτούς που τους τα πούλησαν αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί εμείς στην Ευρώπη δεν είμαστε ικανοί ή να προστατεύσουμε τους πολίτες μας με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ε, χαίρομαι για τη διαδικασία επί παραβάση ε, για τα κράτη-μέλη. Δεν τα, δεν καταλαβαίνω βέβαια όλα, γιατί η Ιταλία, για παράδειγμα, ε, για το θέμα της Ιταλίας ήδη υποτίθεται ότι είναι 300 ευρώ αναπερίπτωση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα φοβήσει τη Fiat ή κάποιον άλλον. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το γιατί. Γιατί αποφασίσατε να εστιάσετε την προσοχή σας στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη και να ξεκινήσετε τη διαδικασία επί παραβάση μόνο για αυτά. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη δεν δρούν, συνεχίζουν να μην δρούν. Ο Γερμανός Υπουργός είπε ότι το να ζητήσουμε, να μην επιβάλλουμε, να ζητήσουμε από τη Volkswagen να επισκευάσει τα αυτοκίνητα αποτελεί αρκετή τιμωρία για την Volkswagen. Αυτό δήλωσε, να ζητήσουμε, το καν να την αναγκάσουμε. Και εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό φτάνει και είναι αρκετό καθόλου τι μπορούμε να κάνουμε να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πολύ πιο ενεργητική δράση από ό,τι το πράττουν τώρα. Και τέλος, ζητήσατε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ να μιλήσει με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε σύνοδο κορυφής για αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το λύσει μόνο η αρμόδια επίτροπος εσείς δηλαδή. Μιλούμε για μια εγγενή λειτουργία της Ευρώπης, τα κράτη-μέλη πολύ απλά δεν συμμορφούνται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ξεκάθαρα και κατάφορα και απολύτως ανοιχτά αρνούνται να συμμορφωθούν. Και εγώ νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εναρκτήρια δήλωση του Προέδρου Γιούγκερ στην έναρξη της επόμενης Συνόδου Κορυφής ή τουλάχιστον η δήλωση του Προέδρου Γιούγκερ στις διμερείς του επαφές με τα κράτη-μέλη. Μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Θα ήθελα να συνεχίσω και εγώ μετά τις ερωτήσεις αυτές που έθεσε ο κύριος Γκερμπράντι, αλλά να δώσω διαφορετική έμφαση σε διαφορετικά ζητήματα. Η επίδελπος μας είπε ότι τίποτα δεν άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες. Εμείς τι ακριβώς όμως κάνουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή και τι ακριβώς έχει κάνει παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τους δύο συνεισηγητές ότι δεν έχουν γίνει ακόμα αρκετά πράγματα. Αν δείτε όμως το σύνολο των διαδικασιών υπαραβάση, όλες αυτές οι ανακοινώσεις, όλες αυτές τις δηλώσεις από πλευράς Ιταλίας και Γερμανίας, δεν μπορούμε να λέμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίσω λίγο περισσότερο από εσά τι εννοείται όταν λέτε ότι τίποτα δεν άλλαξε γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικό και για μας που εργαστήκαμε τόσο σκληρά στα πλαίσια μιας εξεταστικής επιτροπής. Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε δύο εκθέσεις, δεν μπορείτε να λέτε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έπειτα όσον αφορά το agency, τον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση και στη δική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για την πλατφόρμα αυτή που θα πρέπει να δημιουργηθεί έναν οργανισμό, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε, πώς θα συμβάλλουν σε αυτόν τα κράτη-μέλη, ποιος είναι επικεφαλής αυτού του οργανισμού. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να εστιαστούμε στο ότι ε, τα όσα κάνουμε εδώ πέρα θα πρέπει να έχουν και συγκεκριμένες συνέπειες. Εσείς είπατε ότι ε, καταγράφετε όλες αυτές τις συστάσεις επιτροπής μας όσον αφορά την αναδιάρθρωση της όλης προσέγγισής μας. Εγώ προσεγγίζω τα πράγματα όμως λίγο διαφορετικά. Η ειδοποιώς διαφορά της Ευρώπης είναι ότι πολύ συχνά αναλωνόμαστε σε πάρα πολλές συζητήσεις, γίνονται πάρα πολλές ανακοινώσεις και δηλώσεις, αλλά στην πράξη θα θέλουμε να γνωρίζουμε τι θα αλλάξει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε ότι καταγράφετε εσείς και ότι λαμβάνετε δεόντως υπόψη τα όσα λέμε, αλλά θα θέλαμε να δούμε και συγκεκριμένες ε, επιπτώσεις στη συνέχεια, κάποιες βελτιώσεις. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να επιβληθούν επιτέλους. Ποιες βασικές αλλαγές προτίθεστε εσείς να κάνετε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που είναι πολύ σημαντική και για μας και για σας πιστεύω. Συντοπείτε κι εσείς, όπως και εμείς, ότι τα κράτη-μέλη και η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αναλαμβάνουν το ρόλο τους, δεν παίζουν το παιχνίδι και ότι δεν εφαρμόζουν τελικά τους κανόνες. Αυτό προφανώς πρέπει να αλλάξει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό Νομίζω ότι οι συστάσεις και τα δικά μας τα συμπεράσματα, τα οποία θα παρουσιάσουμε στις δύο εκθέσεις μας, της εξαστικής μας αυτής επιτροπής, θα πρέπει πραγματικά να αντιχίσουν πάρα πολύ χειρά προς όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Προλαλήσας σα αναφέρθηκε σε έναν εξάρτητο οργανισμό που θα πρέπει να συσταθεί, προκειμένου η έλεγχη να είναι αμερόληπτη και πιο αποτελεσματική. Αυτή είναι μια πρόταση που πολλές πολιτικές ομάδες υποστηρίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, αλλά και στα πλαίσια της συζήτησης που έλαβε χώρα, αλλά και στα πλαίσια της ψηφοφορίας που θα λάβει χώρα σε λίγο στην ΙΜΚΟ όσον αφορά την έγκριση τύπου. Για τον οργανισμό λοιπόν αυτόν και εσείς το παραδεχθήκατε, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και αν τα κράτη-μέλη ή η αυτοκινητοβιομηχανία δεν τηρούν του κανόνε, αν μη τι άλλο, θα υπάρχει ένα ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίο θα, οποίος θα μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένε αποφάσει. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βλέπω ότι και εσείς εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνείτε με την πρότασή μας αυτή και θα δείτε ότι γίνεται σχετική πρόταση και μνήα στη δική μας την έκθεση. Κυρία Πέτροπε, κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2017 όσον αφορά τα οχήματα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην Ένωση. Ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσει από τα επισκευασμένα αυτοκίνητα της Volkswagen προκειμένου να διασφαλίσει ότι όντως αυτή τη φορά τα οχήματα αυτά τηρούν τους κανόνες και τις ε, προβλεπόμενες προδιαγραφές όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων, ώστε να υπάρχει και έγκριση της KBA. Όσον αφορά τώρα τις οδηγίες αυτές, αναφέρεστε εσείς σε ένα πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο έχει προτείνει και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ακρόση που είχαμε μαζί σας τον Ιανουάριο, είχε γίνει μια κάποια παρουσίαση. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια στοιχεία στο παράρτημα του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι για λόγους αποτελεσματικότητας έχετε βάλει τα στοιχεία αυτά στο παράρτημα και όχι στο διδακτικό του κειμένου. Θα θέλαμε όμως από εσά περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τώρα την τέταρτη δέσμη για τις εκπομπές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης RDE4 υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Και κάτι ακόμα. Το σκάνδαλο Dieselgate ε, προφανώς βρίσκεται ακόμα εξελίξει όπως βλέπετε γιατί έχουμε αποκαλύψεις κάθε μέρα και αφορά και άλλες ε, αυτοκινητοβιομηχανίες και Ευρωπαίους κατασκευαστές. Ως προς αυτό λοιπόν και ως προς ε, την ύποπτη συμπεριφορά πολλών κρατών μελών αλλά και αυτοκινητοβιομηχανιών για τα οξύδια ζώτου και για τα μικροσωματίδια, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ημών, καθώ επίση και μια πιο αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματο για να βελτιωθεί η κοινοτική νομοθεσία. Έχουμε πολλού ε, ευρωσκεπτικιστέ απέναντί μα αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν εμεί να λάβουμε μια πολιτική ευθύνη, να είμαστε γρήγοροι, αποτελεσματικοί και να διασφαλίσουμε ότι η ε, νομοθεσία αυτή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί επεξεργασία όντω θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη και από την αυτοκινητοβιομηχανία υπέρ των Ευρωπαίων καταναλωτών. Συμφωνώ λοιπόν με του δύο συγητέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Ντεσμάγκερ ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με ανησυχεί. πολύ αυτό που είπατε, κυρία Επίτροπε, στην αρχή. Είπατε ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου οι νοοτροπίες, οι στάσεις, ούτε, ε, η στάση των κρατών μελών, η στάση της αυτοκινητομηχανίας. Λέτε ότι πρέπει να κάνετε περισσότερα, αλλά δεν λέτε με ακούλπα. Και επαναλαμβάνω και εγώ το ερώτημα του κυρίου Βαντεκάμπ και θέλω και να το εμβαθύνω. Συμφωνούμε όλοι και λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ομοιόμορφη αντιμετώπιση της αγοράς. Η πρόταση αναθεώρησης της κείμενης νομοθεσίας είναι υπό επεξεργασία. Η Επιτροπή ΕΝΒΙ ε, ψήφισε, έχει σχέδιο γνωμοδότησης στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς επίσης και ένα σημαντικό ερώτημα ήταν η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής, μιας αυτόνομης υπηρεσίας για την παρακολούθηση και την εποπτεία της αγοράς. Και πιστεύω ότι αυτό το αίτημα για τη δημιουργία νέων φορέων, νέων υπηρεσιών πρέπει πάντοτε να εξετάζεται ενδελεχώς και εγώ αυτό το έχω πράξει και πιστεύω ότι ενδείκνυται απολύτως αυτή η υπηρεσία, η σύσταση μιας υπηρεσίας. Έχουμε ανεξάρτητη αρχή για τα σιδηροδρομικά, για τα διαστημικά, για την αεροναυπηγική, αλλά δεν το έχουμε για τις οδικές μεταφορές. Τι πιστεύετε, αξίζει να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία κεντρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα ήταν αυτό πρόοδο. Εγώ πιστεύω πως ναι. Και στη συνέχεια η απόκληση των μετρήσεων εκπομπών στο εργαστήριο και σε συνθήκε ε, πραγματική οδήγηση είναι πολύ μεγάλη. Και αυτή η απόκληση, αυτό το χάσμα το 2016 μεγάλωσε. Ακόμα περισσότερο και θα παραμείνει η απόκληση αυτή ακόμα και μετά τη θέσπιση και υιοθέτηση νέων μεθόδων δοκιμών και ε, εξετάσεων στο εργαστήριο. Ερωτώ λοιπόν, αναγνωρίζετε αυτό το πρόβλημα ε, και τι, τι δράσεις θα αναλάβετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γεφυρώσετε αυτό το χάσμα στις μετρήσεις του εργαστηρίου και στις μετρήσεις σε σύνθηκες πραγματικής οδήγησης. Τι θα γίνει με την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ε, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέτει ε, ορθές πληροφορίες και σωστά στοιχεία και για τη χρήση και για το ύψος των εκπομπών του κάθε οχήματος. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να έχει και πληροφόρηση για το μονοξίδιο του αζότου, για τα πολύ λεπτά και μικρά σωματίδια. Σε μία από τις τροπολογίες που έχω υποβάλει, Προτείνω τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσουν διάλογο με την αυτοκινητοβιομηχανία και να συνάψουν συμφωνίες για το ελάχιστο ε, ύπος επενδύσεων ε, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Συμφωνείτε με αυτή την τροπολογία. Η κυρία Έρνστ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας μας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Χαίρομαι γιατί κάνατε και κριτική. Αυτό χρειάζεται γιατί ε, μας είπαν στις ακροάσεις πράγματα που δεν έστεκαν πολλές φορές. Ε, όλοι παρουσιάζονταν αθώοι ε, έγιναν ε, ε, προσπάθειες προβολής συμφερόντων, όλα τα είδαμε, όμως δεν μάθαμε όλα αυτά που θέλαμε. Και αυτό είναι και ένα μειονέκτημα της Επιτροπής μας που ήθελε όλα τα έγγραφα να τα λαμβάνει έγκαιρα πολλές φορές ε, δημιουργήθηκαν προβλήματα για τα οποία δεν ήταν υπέτεια η Επιτροπή μας. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα που χρειάζονται για τις εξεταστικές επιτροπές ε, και στο μέλλον. Ο ε, ε, επικεφαλής πίσω, ε, ακούσαμε χθες τις ειδήσει, κατηγορεί τους μεγαλομετόχους για το γεγονός ότι υπάρχουν παρατυπίες και βλέπουμε ε, στενή διαπλοκή πολιτικής και οικονομίας, πράγμα το οποίο δεν ε, είναι θετικό για την δική μας την προσπάθεια. Η εστίαση η δική σας κυρία Επίτροπε είναι πολύ σημαντική γιατί μιλήσατε για ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Ε, εμείς ε, ε κάναμε μια σοβαρή δουλειά ε, προσπαθήσαμε δηλαδή να εργαστούμε σοβαρά. Αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί με βάση τις συστάσεις που θα προκύψουν από την έκθεση που θα ε, υποβληθεί και να ε, εξαχθούν συμπεράσματα. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει δηλαδή να υλοποιηθούν. Επίσης, τι γίνεται με την δουλειά των λόμπι. Αναφέρομαι στο άρθρο 6 του σχεδίου έκθεσης που λέει ότι ε, περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη της ε, ε, Επιτροπής RDV-LD V αποτελείται από μέλη της, του κλάδου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εκπροσώπους των λόμπι. Θα πρέπει να είναι, το θεωρήσουμε αυτό πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες επιτροπές ή όχι. Επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα ψήφου καλό είναι να μας πείτε ορισμένα πράγματα για τους εκπροσώπους του λόμπι, γιατί πολλοί συνέβαλαν στην ε, συναγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Επίσης, θέλουμε ό,τι αποφασιστεί το πακέτο RDE και όλα τα σχετικά θα πρέπει να ε, είναι αυστηρά, θα πρέπει να υπάρχει δημόσια βάση δεδομένων η οποία να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών RD. Αυτό είναι κατεπήγον και θα ήθελα να μου πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε την ε, άρνηση των κρατών μελών να συνεργαστούν. Ε, εκτός από τη διαδικασία επιπαραβάση υπάρχουν και άλλα μέσα στη διάθεσή σας για να πείσετε τα κράτη-μέλη, να ασκήσετε πίεση σε αυτά. Τα κράτη-μέλη δεν είναι ε, όλα ενθουσιώδη, αλλά ούτε και οι, όλες οι πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία. Επίσης, τέλος, θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό η Κομισιόν θα ε, ε, θεσμοθετήσει μηχανισμούς ασφαλείας, ούτως ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα και να προλαμβάνονται, ούτως ώστε να αποφευχθούν παρόμοια σκάνδαλα. Ε, μην ξεχάσω και τα ε, μικροσωματίδια, πρέπει και αυτό να ε, συμπεριληφθεί. Η εμπιστοσύνη βέβαια ε, κερδίζεται όταν κανείς είναι συνεπής στην δράση του. Θα πρέπει να δούμε ε, λοιπόν και τα κράτη-μέλη, το ρόλο που έπαιξαν, αλλά και το ρόλο της Κομισιόν, γιατί ε, πολλές φορές αποκρύφτηκαν πράγματα, ε, πράγμα που έδειξε και η ακρόαση με προηγούμενους επιτρόπους, πρώην επιτρόπους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις σαφείς αυτές δηλώσεις που κάνατε και συμμερίζομαι και εγώ την έκπληξη ε, πολλών συναδέλφων. Δυστυχώ όμω να γνωρίσουμε όλο και περισσότερο ότι η στάση του Συμβουλίου δεν έχει ουσιαστικά τροποποιηθεί πάρα πολύ. Δεν μπορούμε εμεί όμω να μείνουμε μόνο σε αυτό το συμπέρασμα και προφανώ υπάρχει ένα ρόλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό θα ήθελα λοιπόν να εστιαστώ αναφερόμενος στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες όσον αφορά τα συστήματα αναστολής όπου έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ πλέον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ μπορούν να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν αυτά τα συστήματα, οι διατάξει αναστολή. Αυτή τη στιγμή συνδυάζουμε πολλά στοιχεία που μα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δούμε τι οδηγίε αυτέ, αυτέ τι καθυντήριε γραμμέ, μα κάνει ακόμα εντύπωση όταν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει το πρωτογενέ δίκαιο. Αν δούμε τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λάβαμε ως Εξεταστική Επιτροπή, την Καλέχα για παράδειγμα, οι ε, φυσιολογικές συνθήκες ε, λειτουργίας και οδήγησης δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κύκλο δοκιμών. Λέγεται λοιπόν ότι ο νόμος είναι σαφής και ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα θα πρέπει σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης να πληρούν και να τηρούν τα πρότυπα αυτά και όχι μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες. Αν διαβάσετε όμως οδηγίες και τις κατευθύνες γραμμές για τα συστήματα αναστολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει για παράδειγμα ότι αν κάνουμε δοκιμές με σύστημα RDE, τότε υπάρχουν ακόμα οχήματα τα οποία μπορούν να εκπέμπουν διπλάσιο ή και πενταπλάσιο ποσοστό ρήπων από αυτό το οποίο προβλέπετε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνάδει καθόλου με το συντελεστή συμμόρφωση που εσεί οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνατε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να ανέχεστε ότι στα πλαίσια των δοκιμών RD μπορείτε να έχετε πενταπλάσια εκπομπή ρήπων από την προβλεπόμενη. Και ότι στην περίπτωση αυτή λέτε ότι μπορεί τότε να φανεί ότι όντω χρησιμοποιείται από ένα όχημα σύστημα αναστολή. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να μπορούμε να εντοπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Δεν προβλέπεται επίση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Λέτε ότι μπορεί ένα όχημα ξαφνικά να εκπέμπει πεταπλάσια ποσότητα ρήπων από την επιτρεπόμενη και μόνο στην περίπτωση αυτή μπορείτε εσείς να αρχίσετε κάποιες έρευνες για να δείτε τελικά αν το συγκεκριμένο αυτό όχημα μπορεί να περιέχει ένα σύστημα αναστολή. Επίσης, με μια πολύ μικρή αλλαγή που μπορεί να γίνει σε επίπεδο κινητήρων, τότε μπορεί και ένα αυτοκίνητο να αρχίσει να εκπέμπει το σωστό ποσοστό ρήπων. Ξέρετε ότι γίνονται και πολλές εθνικές έρευνες. Στη Γαλλία έγινε μία δοκιμή της κατηγορίας 1, στα πλαίσια της οποίας γίνανε και πολλά, πολλά και σημαντικά πράγματα. Στην γαλλική λοιπόν αυτή η έρευνα είδαμε ότι η Αλφα Ρωμαίο με μικρές μόνο αλλαγές στις δοκιμές αυτές πάλι εκπέμπει 399% περισσότερο. Η Ford το ίδιο, η Fiat το ίδιο, η Nissan πάνω από 450%, η Opel σχεδόν 200%, η Renault 250%, η Volvo 160%. Εσείς ε, στις οδηγίες σας έχετε θέσει ανώτατο όριο. Είπατε ότι δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε το 10%. Όλα αυτά τα οχήματα στα οποία αναφέρθηκα, ουσιαστικά συνδυάζουμε αυτή τη στιγμή τις δικές σας κατευθύνες γραμμές με τις εθνικές έρευνες, βλέπουμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε όλες αυτές τις δοκιμές έχουν υπερβεί κατά πολύ τα οχήματα αυτά τις ε, προβλεπόμενες ε, εκπομπές και λέτε ότι στις περιπτώσεις αυτές καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια απαγορευμένη διάταξη αναστολής χρησιμοποιείται. Το λέτε και εσείς λοιπόν στις δικές κατητήριες γραμμές, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ουσιαστικά έχουμε εντοπίσει συστήματα αναστολής και έχουμε και ένα νομικό σημείο μας στη συνέχεια, στο οποίο λέει ότι αν εντοπίσουμε τέτοιες απαγορευμένες διατάξεις αναστολής, οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να αποσύρουν, να ανακαλέσουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία περίπτωση και σε κανένα κράτος μέλος. Αν τα συνδυάσουμε λοιπόν όλα αυτά καταλήγουμε στο εξή απλό συμπέρασμα. Πολλά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή δεν συμμορφώνονται με το νοσιακό δίκαιο. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μόνο πράγμα μπορεί να κάνει, να κινήσει διαδικασίε επί παραβάση. Και δεν αναφέρομαι σε διαδικασίες παραβάση όσον αφορά τον ορισμό και τον καθορισμό των συστημάτων αναστολή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται συστήματα αναστολή και εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα. Η ενωσιακή νομοθεσία λέει ότι απαγορεύονται τα συστήματα αναστολή. Λέγεται αυτό ρητά στην ενωσιακή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα και επ' αυτό να κινήσει διαδικασίε ε, επί παραβάση και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα οχήματα αυτά δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν καν στους ευρωπαϊκούς δρόμους και προφανώς δεν θα πρέπει να μολύνουν και δεν θα πρέπει να έχουν καν πιστοποιητικό συμμόρφωση όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Το ενιαίο κέντρο ερευνών, το κοινό κέντρο ερευνών και η γαλλική πλευρά επίσης κάνανε δοκιμές όπως σας είπα στα πλαίσια της κατηγορίας 1. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες δοκιμές στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας. Γιατί βλέπετε ότι τόσο περισσότερο κάνουμε έρευνες, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν συστήματα αναστολής. Ας πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία έχει το λόγο. Η κυρία λόγο. ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την διαφωτιστική αυτή ανάλυση του bass Out, ουσιαστικά βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι η φυστάμενη κατάσταση είναι πολύ πιο ανησυχητική, πολύ περισσότερο ανησυχητική από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τις ε, γερμανικές και ιταλικές αρχές σε σχέση με τις έρευνες που έχουν γίνει για την ύπαρξη συστημάτων αναστολής. Θα ήθελα να καταλάβω ποιος είναι ο ρόλος ο δικό σας και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των ερευνών αυτών και της αντιπαράθεσης που έχει προκύψει ανάμεσα στις γερμανικές και τις ιταλικές αρχές. Εσείς προσπαθείτε να διευκολύνετε την ανταλλαγή απόψε και τον διάλογο ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη ή μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις ανεξελίξει έρευνες προκειμένου να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένα πορίσματα πέρα από αυτά που έχουμε δηλαδή όσον αφορά την χρησιμοποίηση διατάξεων αναστολής και στην αντίθετη περίπτωση όταν κλείσει η δικαστική αυτή διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες και εφόσον κάθε χώρα μείνει οχυρωμένη στη δική της τη θέση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση αυτή. Ο Ιταλός Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Ντελερίο, μιλώντας σε μια ακρόαση του Ιταλικού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στο ότι θα κλείσει όλη η υπόθεση αυτή με έναν τρόπο αισιόδοξο κατά αυτόν. Νομίζουμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις ε, όσον αφορά την υπόθεση της Fiat. Η Fiat έχει πει ότι ε, εθελοντικά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία τροποποίησης του software που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Συμφωνείτε κι εσείς ότι όντως θα κλείσει αισιόδοξα η όλη αυτή η ιστορία και το γεγονός ότι ε, η Fiat έχει αρχίσει να κάνει κάποιες αλλαγές όσον αφορά το σύστημα των αυτοκινητωμάτων και συγκεκριμένα των αυτοκινήτων με συγχωρείτε και του λογισμικού τους. Είναι για σας κάτι το οποίο είναι θετικό. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όντως θετικά την όλη αυτή η ιστορία και εν τέλει μήπως ε, όλοι θα βγουν αλόβητοι από την ιστορία αυτή καθότι δεν θα επιρρύψουμε ευθύνε σε κανέναν. Και τα λέω όλα αυτά σε σχέση με αυτά που είπατε και στην αρχική σας παρέμβαση. Είπατε ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση όσον αφορά τη στάση των κρατών μελών και ότι δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή κάποια θετική πολιτική βούληση προκειμένου να συνεργαστούν περισσότερο με εμά. Μπορείτε να σχολιάσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους συναδέλφους. Η κυρία Γκροστέτ έχει δηλώσει ότι θέλει το λόγο. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο να μου το πείτε τώρα. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε για αυτή τη συζήτηση η οποία είναι όντως σημαντική τη στιγμή που συντάσσουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής. Δεν θα επανέλθω στα ζητήματα που έχουν ήδη θίξει διάφοροι συνάδελφοι. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ξαναμιλήσω για τους καταναλωτές και την ε, απόγνωση στην οποία βρίσκονται σήμερα, διότι ε, θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο και αναρωτιούνται. Αλήθεια μας λένε. Από ό,τι φαίνεται οι πωλήσει αυτοκινήτων diesel έχουν μειωθεί πάρα πολύ ε, φέτος. Πώς βλέπετε το μέλλον. Μας αφορά όλους το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ένας κλάδος της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας πολύ, σημαντική, σημαντικός Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το μέρισμα μεταξύ ε, βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων, υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη και οχημάτων που κινούνται με άζωτο και διάφορες άλλες εναλλακτικές μορφές. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να μην υπάρξει ένα τεράστιο οικονομικό σοκ στον κλάδο ξαφνικά. Η αυτοκινητοβιομηχανία ε, κάνει έρευνα, ε, αναπτύσσει το ντίζελ με νέες τεχνολογίες καλύτερες. Τι πιστεύετε, εάν υπάρχουν ενδιαφέρουσες τεχνολογίες στον τομέα του ντίζελ, θα τις στηρίζατε ή όχι. Θέλουμε να μάθουμε. Πολλοί είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανωθεί διαφορετικά, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα και πρέπει να ε, βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Διεθνούς και Ερευνητικού Κέντρου και των αρμοδίων γενικών διευθύνσεων. Είδαμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν ε, κυκλοφορούσαν ε, σωστά. Πώς θα δράσετε για να υπάρχει απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών στο μέλλον. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης μιας εργασίας, μιας δουλειάς, η οποία χρησιμεύσει στην ανάδειξη των εξή συμπερασμάτων. Ότι δηλαδή δεν, ε, ότι απέτυχαν οι έλεγχοι και δεν τηρήθηκαν οι συστάσεις οι κατευθυντηρίες γραμμές και τελικά είχαμε μια περίπτωση απάτης, εξαπάτησης που έπληξε άμεσα τους χρήστες, τους καταναλωτές και πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία ήταν επιχείρηση ή επιχειρήσεις που ουσιαστικά κορόιδευαν τους κανόνες για να επιτύχουν στόχους απορριπταίους. Επομένως η εργασία και η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν ε, μια δουλειά του να απαιτήσει να αναλάβουν την ευθύνη τους οι ένοχοι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Δουλειά της Κομισιόν ήταν να δείξει το δρόμο προς τα που πρέπει να κινηθούμε να ε, ε, δώσει τους προσανατολισμούς έτσι ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μην ξανασημειωθούν ποτέ. Σήμερα έχουμε τις ε, εγγυήσεις ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει. Τα συμπεράσματα χρησιμεύουν στο να πούμε ότι εδώ βάζουμε τη τελευταία τελεία σε μια ιστορία η οποία δεν θα ξαναυποθεί και δεν θα ξανασυμβεί. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την εγγύηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη, είναι υποχρεωμένη να μας προσφέρει εγγυήσει ότι μια τέτοια κατάσταση δεν θα επαναληφθεί γιατί αλλιώς δεν είμαστε αξιόπιστοι. Στην διάσκεψη των Παρισίων για, τον, για το κλίμα, θέσαμε στόχους εξαιρετικά φιλόδοξους. Δεν είμαστε αξιόπιστοι όταν πηγαίνουμε στο Παρίσι να θέτουμε και να υπογράφουμε τέτοιους στόχους και μετά να μην αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις στην πράξη. Χάνουμε έτσι την αξιοπιστία μας. Πρέπει να έχουμε εργαλεία που θα υποχρεώνουν τα κρατη να τηρούν τις αποφάσεις. Χρειάζεται ε, αποφασιστικότητα, χρειάζεται πολιτικό θάρρος. Και μιλώ μόνο για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι μιλώ και εξ ονόματος ε, πολλών συναδέλφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να σας στηρίξει όταν θα πάρετε αυτές τις αποφάσεις, παρόλο που οι αποφάσεις αυτές κοστίζουν και είναι, δαπανηρές. Θέλουμε να αποφύγουμε να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και αυτό έχει κόστος και είμαστε έτοιμοι να το αναλάβουμε. Άλλωστε, το κόστος προστασίας του κλίματος και της υγείας των ανθρώπων δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Και γι' αυτό αξίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ζητούμε να είστε πιο αποφασιστικοί, να, να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση με πιο αποφασιστικό τρόπο, με βάση τις αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει. Ο κύριος Ενρίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σχόλια Καταρχάς, να μην επαναλάβω το γενικότερο, τη γενικότερη αίσθηση των συναδέλφων, τη συμμερίζομαι απολύτως. Να πω όμως ότι σε αυτή την υπόθεση φαίνεται ότι όλη η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδόν εμπλέκεται. Το κέντρο ελέγχων ε, δεχόταν επιστημονικά μια μέθοδο η οποία είχε πάρα πολλά κενά. Δηλαδή όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας τελικά αποδείχθηκαν αδύναμοι, με μικρή επιμέλεια, δεν έκαναν το δέον γενέστε. Συμφωνώ λοιπόν με ε, την πρόταση των συναδέλφων να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει με ε, σωστές ε, προϋποθέσεις και σωστούς όρους όλους αυτούς τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή την θλιβερή υπόθεση. Αν δούμε όμως το πώς ξεκίνησαν τα πράγματα από την αρχή, ε, θα θυμηθούμε το εξή. Μετά από τη δημιουργία διαφόρων τεχνικών επιτροπών, ομάδων εργασίας κτλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε κανόνες στήρισης εκπομπών για μονοξίδιο ε, του αζότου, διοξίδιο του άνθρακα κτλ. Και καθορίστηκαν τότε, τότε τα κατόφλια που παρόλα αυτά δεν τηρήθηκαν και ποτέ. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω όμως είναι το εξής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό ποιες συνθήκες έγιναν από τους αρμόδιους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Γιατί το κατόφλι των εκπομπών και στη συνέχεια οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν προέκυψε πώς. Ε, έγιναν ομάδες εργασίας που κατέληξαν σε κάποια νούμερα τα οποία τελικά ήταν κενά, δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επομένω, πώ κατέληξαν σε αυτά τα νούμερα που δεν υπήρχαν, αφού τελικά φάνηκε ότι τα ξεπερνούν τα αυτοκίνητα κατά πέντε φορέ. Δηλαδή, οι κανονιστικές και νομοθετικές προτάσεις που είχαν γίνει τότε δεν ανταποκρίνονταν σε καμία τεχνική πραγματικότητα. Και, ούτε, και μετά ε, ε βεβαίως αποδείχθηκαν και παρανομούσες οι, οι επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στους ελέγχους. Άρα, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στις προτάσεις της ήξεραν, είχαν ιδέα ε, ότι οι δικές τους προτάσεις πόρα απέχουν από την πραγματικότητα, είναι από άλλο κόσμο ή ξέρανε ότι ό,τι νούμερο και να, βάλανε, να βάζανε στα κατόφλια και στις εκπομπές δεν θα είχε καμία σημασία γιατί ο κλάδος θα το παραβίαζε. Ευχαριστούμε. Στρεφόμαστε τώρα στην κυρία Επίτροπο, η οποία έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, Αν θέλετε να δώσω λεπτομερείς απαντήσεις στις λεπτομέρειες ερωτήσεις σας, τότε προτιμούσα να το κάνω αυτό γραπτός. Καλύτερα να απαντήσω εν γέννη στις παρατηρήσεις σας εδώ εν ώψη της Επιτροπής σας. Ας ξεκινήσω λίγο με το ζήτημα των αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο τέθη και θα ήθελα να μαθοποιήσω κάπως απαντήσεις που θα σας δώσω στη συνέχεια. Όπως θα ακούσατε ήδη πολλές φορές, πραγματικά ασκούσα πίεση και προσπαθούσα να πείσω την Volkswagen ε, θελουσίως να αποζημιώσει τους Ευρωπαίους πολίτες, τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Στα πλαίσια της ενωσιακής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσία επιβολής ε, της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Μαζί με την Επίτροπο Γιούρεβα, η οποία και αυτή συζήτα πάρα πολύ με τα κράτη-μέλη και τις ενώσεις των καταναλωτών, προσπαθούμε από κοινού να επιβάλλουμε την ενωσιακή νομοθεσία με διαφορετικούς τρόπους σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα κολλάνε σε αυτό το οποίο είπατε πάρα πολύ από εσά, ότι δεν είχαμε την απαραίτητη συμβολή τόσο των κρατών μελών όσο και τη αυτοκινητοβιομηχανία. Το ζήτημα των αποζημιώσεων χρειάστηκε να το συζητήσω πάρα πολλέ φορέ με τη Volkswagen και πραγματικά είναι απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αυτή και άλλες εταιρείες αντιμετωπίζουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα συνεχίσω να σκώ πίεση, διότι θα με βοηθήσει πιστεύω πάρα πολύ και η δική σας η έκθεση στο εγχείρημά μου αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική νομοθεσία, αλλά είναι απαράδεκτο θα έλεγα να μπορούμε να ανεχόμαστε ένα σύστημα απλών ανακλήσεων χωρίς να προβλέπονται άμεσες αποζημιώσεις για τους ε, Ευρωπαίους ε, καταναλωτέ που έχουν ζημιωθεί. Θα ήθελα να πω ότι στην Ιταλία οι αποζημιώσει ήταν 300 ευρώ, 300.000 ευρώ ένα αυτοκίνητο. 300 με συγχωρείτε ευρώ ένα αυτοκίνητο. Και όπως είπατε και εσείς δεν ήταν πολύ ψηλό το ποσό αυτό, συμφωνώ. Κάτι άλλο που σας προκάλεσε εντύπωση, το αναφέρατε πολύ, όντως σε καθημερινή βάση συζητούσαμε το ζήτημα αυτό και με την αυτοκινητοβιομηχανία και με τα κράτη-μέλη. Ήδη χθε προχθές κάναμε μια άλλη συζήτηση τέτοια και θα έλεγα ότι η πραγματική φύση αντιμετώπιση από την αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει τροποποιηθεί. Αρνούνται όλα αυτά τα γεγονότα και έχετε δίκιο περισσότεροι όταν λέτε ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά δεν κατάφεραν να επιβάλλουν νομοθεσία. Ένα είναι αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως πολύ σωστά το θίξατε. Έχω καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες και με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι έκανα κάθε τι το δυνατό. Κάθε τι το δυνατό. Έκανα ό,τι μπορούσα. Τρία πράγματα. Ένα νέο σύστημα έγκριση τύπου καταρχά. Γιατί τα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε μέχρι στιγμή είναι πάρα πολύ περιορισμένα όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής της νομοθεσίας. Στην προηγούμενη παρέμβασή μου εδώ στην Επιτροπή σας, κατά τη διάρκεια της Σας είχα πει ότι θέλουμε μια πολύ καλή βάση δεδομένων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Το κάναμε το Δεκέμβριο κατά 7 κρατών μελών και είχαμε μια πολύ καλή βάση δεδομένων. Η καταλεκτική ημερομηνία για να λάβουμε απαντήσεις από τα κράτη-μέλη είναι σήμερα, επομένως θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τώρα τις απαντήσεις τους. Δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, Πάντω πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα νέο γύρο διαδικασιών παραβάση του επόμενου μήνε. Ξέρετε ότι όμω τα μέσα αυτά που έχουμε είναι πολύ περιορισμένα. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα έγκριση τύπου, το συντομότερο δυνατό. Αυτό επίγει. Θα πρέπει να αλλάξουμε το σύνολο του συστήματο, του ελέγχου των εκπομπών ρήπων και να μπορούμε επίση να ελέγχουμε και τι ίδιε τι αρχές έγκρισης τύπου. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε έναν εξάρτητο οργανισμό. Θα έλεγα ότι στο 90% των συστάσεών σας υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα σημείο όμως επί του οποίου διαφέρει η άποψή μου από τη δική σας. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε έναν ξεχωριστό ευρωπαϊκό οργανισμό. όπως η αντίστοιχη EPA των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε ανταυτού είναι ένα σύστημα επίβλεψης της αγοράς που να είναι ανεξάρτητο από την επίβλεψη που κάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Γιατί όπως σας είπα στην αρχική μου παρέμβαση, τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν προσκολλημένα στην ιδέα ότι είναι τα μόνα ηθήνοντα, τα μόνα υπεύθυνα για την ε, μέτρηση των εκπομπών ρήπων στα αυτοκίνητα. Δεν δεχόντουσαν ουσιαστικά νουθεσίες ή παρεμβάσεις από κανέναν άλλον οργανισμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα νέο μηχανισμό επιτήρησης αγοράς που θα είναι αποτελεσματικός. Θα πρέπει επίσης να καταβληθούν και κάποιες χρηματοδοτικές προσπάθειες. Όπως το είπα και σε προηγούμενη μου παρέμβαση στην Επιτροπή σας, ακριβώς επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ακριβώς επειδή το κόστος είναι πολύ μεγάλο, ακριβώς επειδή οι δημοσιονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές, η εναλλακτική ενός κεντρικού ευρωπαϊκού οργανισμού δεν επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένω να είναι το μόνο σημείο επί του οποίου διαφέρουν οι απόψεις μας. Υπάρχει ταύτιση όμως απόψεων σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Ετέθηκε ένα ερώτημα όσον αφορά την θέση του κυρίου Γιούνκερ επί όλων αυτών. Προφανώ καταλαβαίνετε ότι συλλογικά ο σώμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνουμε την κίνηση διαδικασιών παραβάση. Είναι ενήμερος για όλε αυτές τι περιπτώσει ο πρόεδρο Γιούνκερ. και νομίζω ότι ε, έχει έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου για να δούμε τελικά πώς θα επέμβει το Συμβούλιο. Και θα θέλαμε προφανώς να έχουμε και μία παρέμβαση του Συμβουλίου εν προκειμένου. Είμαι σε καθημερινή επαφή ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα κράτη-μέλη και με τον κλάδο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζομαι τη δική σας την υποστήριξη γιατί θεωρώ ότι ακόμα προσπαθούν να καθυστερήσουν την όλη διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το ζήτημα αυτό. Ξέρω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά τεχνικά δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε, αλλά δεν είμαι υπέρ της προσέγγισης αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι ε, δεν πρόκειται να σημειώσουμε πρόοδο καθόλου με τα οικολογικά αυτοκίνητα, με τα αυτοκίνητα που θα έχουν μηδενικές εκπομπές, αν δεν καταφέρουμε πρώτα να έχουμε ένα νέο σύστημα έγκρισης τύπου. Αν δεν καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτό το νέο σύστημα έγκρισης τύπου, μένουμε εγκλωβισμένοι στην υφιστάμενη κατάσταση. Και το μόνο το οποίο θα έχουμε θα είναι παραβάση παραβάσεων και τίποτα άλλο. Το σύστημα αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εξαλείψει οποιοδήποτε φαινόμενο παράβαση στο μέλλον, αλλά αν μη τι άλλο έχουμε ένα νέο σύστημα έγκρισης τύπου, θα περιορίσουμε πάρα πολύ τα αρνητικά αυτά φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οδηγίες τι οποίε εκδώσαμε. Στο παρελθόν Κανένα κράτος μέλος δεν ζητούσε οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο νόμος είναι ξεκάθαρο. Τα συστήματα αναστολή είναι παράνομα στην Ευρώπη. Η χρήση του είναι παράνομη. Το συζητήσαμε όμω αυτό και στο παρελθόν και σας είχα πει τότε ότι θα προχωρούσε με κατευθυντήρες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εργαλείο αυτό απευθύνεται κυρίως προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορούν να κάνουν πιο σωστές αξιολογήσεις. Ας αποσαφηνίσουμε λίγο τα πράγματα. Όλα αυτά αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην υφιστάμενη νομοθεσία τα κράτη-μέλη είναι τα αρμόδια για τις αξιολογήσεις των εκπομπών ρήπων. Εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο πράξαμε τελικά. Να δημοσιεύσουμε κατευθύντηρες γραμμές. Ελπίζουμε ότι τις οδηγίες αυτές θα τις ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό ζήτημα είναι να έχουμε τη δική σας την υποστήριξη για να έχουμε ένα νέο σύστημα RDE, να έχουμε καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και νέα μέτρα έγκρισης τύπου. Ένα νέο σύστημα έγκρισης τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε στους τρεις αυτούς τομείς, θα σημειώσουμε πολύ σημαντική πρόοδο. Φέτος και στα πλαίσια της υψηλόβαθμης ομάδας με ορίζοντα το 2030 θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή πόσα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές ή εντελώς οικολογικά αυτοκίνητα ή αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν μέχρι το 2030 στους δρόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας απασχολεί σε καθημερινή βάση και με τους εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και κάθε μήνα βλέπουμε ότι το ποσοστό των οχημάτων αυτών όλο και αυξάνεται. Άρα και ο ίδιος ο κλάδος πρέπει να προετοιμαστεί για τη νέα αυτή γενιά αυτοκινήτων και ήδη χθε απευθυνόμενοι σε εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας τους είπα ότι μάλλον έχει έρθει πλέον ο καιρός να αρχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες κυρίως μέσω των ανθρωπίνων πόρων μας και μέσω της χρηματοδότησης πλέον που δίνουμε προς τη νέα αυτή γενιά αυτοκινήτων και να μην επικεντρωνόμαστε πλέον τόσο πολύ ή να μην επενδύουμε πλέον τόσο πολύ σε διζελοκίνητα αυτοκίνητα ή σε αυτοκίνητα παλαιότερης γενιάς. Το ζήτημα αυτό το συζητάμε εδώ και 18 μήνες βέβαια και ολοκληρώνω στο σημείο αυτό πάλι και ως προς αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ θεαματική αλλαγή, αν θέλετε, στη σάση που διατηρεί τόσο η αυτοκινητοβιομηχανία και όσο ε, και τα κράτη-μέλη τα ίδια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, ότι το σκάνδαλο αυτό ήταν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα που χρειάζεται να επενδοποιήσουμε στην Ευρώπη. Θα περιμέναμε λοιπόν μια διαφορετική στάση από τα κράτη-μέλη και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν είπατε τίποτα για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τις διατάξεις αναστολής. Δεν... συμφωνώ μαζί σας ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, εφήρμοσαν την ενωσιακή νομοθεσία και έχουμε κάνει πιο αυστηρή την νομοθεσία από το Μάιο του 2016. Οι κατασκευαστές ε, παρουσίασαν τις στρατηγικές για τις εκπομπές που πρέπει να αξιολογηθούν από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ήταν αυστηρή η κατευθυντήρια γραμμή που τους δώσαμε. τα κράτη-μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τις στρατηγικές εκπομπών τους. Δεν θυμάμαι ή άλλο συγκεκριμένο ρωτήσε. Είπατε ότι δεν συμμορφώθηκαν με την ενωσιακή νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, δεν ε, συμμορφώθηκαν. Δηλαδή ακόμα κυκλοφορούν. Αν δεν συμμορφούνται κανείς, θα πρέπει να αποσυρθούν τα οχήματα. Είναι σαφές το νομικό σημείωμα. Ε, δεν συμμορφώνονται, ε, δεν υπάρχει συμμόρφωση. Θα κινηθεί η διαδικασία επί παραβάση στις χώρες αυτές. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισα αυτό, ναι. Είπατε μπορεί. Αν λέτε όμως ότι δεν συμμορφούνται, τότε πρόκειται για παράβαση και πρέπει να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάση. Βεβαίως, είπα, όπως έγινε με τι 7 παραβάσει το Δεκέμβρη, πρέπει να έχουμε πλήρη, πλήρη δεδομένα, όλε τι τεχνικέ λεπτομέρειε και πρόσθεσα ότι είμαι βεβαία ότι και πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Θα, τις, τους επόμενους μήνες θα κινηθούν οι επόμενες διαδικασίες επί παραβάση. Η κυρία Έρνς, όχι άλλη ερώτηση όμως. Εγώ ε, ρώτησα κάτι για τα λόμπι. και πώς αντιμετωπίζονται οι οργανώσεις τους το απαντήσατε αυτό και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό επηρεάζει τη σύνθεση πολλών σημαντικών επιτροπών. Ε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε συναγάγει συμπεράσματα σχετικά. Ε, τα λόμπι βέβαια είναι ένα γενικότερο θέμα για το Κοινοβούλιο. Να προσπαθήσω να απαντήσω, γραπτός όμως. Γιατί αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το βλέπω αυτό. Και βλέπω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία με τα λόμπι της επηρεάζει και κυβερνήσει των κρατών μελών. Αλλά θα κοιτάξω να δώσω γραπτός περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, ναι, είναι γενικότερο το πρόβλημα. Υπάρχουν ακόμα πολλές, πολλά ανοιχτά ερωτήματα, συμφωνώ. Πολύ ε, θα ήθελα να επανέλθουν. Έχουμε όμως τη συζήτηση για την έκθεση. Εμάς καθήκον μας είναι να στηρίξουμε την Κομισιόν, να είναι πολύ ε, δυναμική, αυστηρή σε αυτά τα θέματα. Αυτός είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη, αυτή θα είναι, όχι, ε, θα, θα είναι η πρώτη τελευταία μας συνάντηση. Μετά θα επιστρέψουμε στις Επιτροπές και θα φροντίσουμε να υιοθετήσει η ΙΜΚΟ τις συστάσεις μας. Διαδικαστικά, ναι, διαδικαστικό κυρία Πρόεδρε. Μέχρι τις 12.30 συνεδριάζουμε και είναι 10 και Δύο ώρες χρειαζόμαστε για τη συζήτηση των τροπολογιών, δεν νομίζω. Ας κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων στην κυρία Πίτροπο, αν το δεχτείτε παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, με ένα λεπτό στο κάθε μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διατυπώσει το ερώτημά του, γιατί εγώ δεν έλαβα κανένα, καμία απάντηση στα ερώτηματά μου. Είμαστε εδώ υποτίθεται για να ανταλλάξουμε απόψεις. Η πρόεδρος. Ε, το καταλαβαίνω και είμαστε πασίγνωστοι για τις μεθόδους ακροασής μας. Είναι κάπως περίεργο να τέθουν τόσα πολλά ερωτήματα τώρα, αλλά η κυρία Επίτροπος πρέπει να πάει σε άλλη επιτροπή τώρα. Ας τις υποβάλουμε ερωτήσεις γραπτός. Ας έχουμε έναν κύριο γραπτών ερωτήσεων και απαντήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν συμφωνείτε όλοι, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Επίτροπο. Okay, Με um, uh, τη συνάδελφοι, γραπτός λοιπόν μπορούμε να υποβάλουμε περισσότερες ερωτήσεις στην Επίτροπο και δεν ολοκληρώνεται εδώ πέρα η διαδικασία βέβαια. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τρίτο, πέμπτο μάλλον σημείο της ημερήσιας διάταξης, για να μακριβείς σχέδιο έκθεση σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη συνέχεια έχουμε και το σχέδιο συστάσεων εν συνεχεία της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεων εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουμε δύο εξαιρετικούς συζητητές, στους οποίους θα ήθελα να δώσω το λόγο, στον κύριο Γκιζέκε δηλαδή και στον κύριο Γκερμπράντι, και θα ακούσουμε στη συνέχεια τους σκιώδεις συγητές και μπορούμε να κάνουμε έπειτα μια συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη. Κύριε Γκιζέκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία που μέχρι τώρα έκανε εξαιρετική δουλειά και μας υποστήριξε πάρα πολύ σε όλες τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Γκερμπράντι και όλους τους σκιώδεις για την επικοδομητική δουλειά. Με την επικοδομητική δουλειά όλων των ομάδων καταλήξαμε σε ένα πραγματολογικό κομμάτι αντικειμενικό, σωστό. Οι ακροάσεις ε, επιδέχονταν πολλές φορές διαφορετικές ερμηνείες. όλα αυτά όμως μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Ε, θα ήθελα να συνεχίσουμε τις συμβιβαστικές ε, διαδικασίες. Ε, έχουμε, είχαμε 205 και 181 τροπολογίες ε, ε, στο σχέδιο έκθεσης και στις συστάσεις. Ε, είχαν τεχνικά προβλήματα για τις συμβιβαστικές, μεταφραστικά προβλήματα, ακόμα στα γερμανικά, τη μητρική μου γλώσσα δεν υπάρχουν οι τροπολογίες, πρέπει να δουλέψουμε με τα αγγλικά, καμιά φορά τα γαλλικά και τα ιταλικά, δεν διευκολύνει τη δουλειά μας, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγητές. Τώρα, έχουμε κάποιες διαφορές. Υπάρχουν εννέα συμβιβαστικέ και οχτώ αντίστοιχα για την έκθεση και τις συστάσεις. Θα συζητήσουμε και στο Στρασβούργο. Από την άποψη του ΕΛΚ ε, υπάρχουν ορισμένες προτεραιότητες που δεν πρέπει να ε, παραμεριστούν. Ε, πρόκειται για τεχνολογία του μέλλοντος. Ήδη μπορούμε να έχουμε οριακέ τιμές ε, στα αντιζελοκίνητα, θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες που υπάρχουν. Τότε γίνεται. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ε, τα, το ντίζελ για τελογικούς λόγους. Τώρα, για το conformity factor και την νομοθεσία RDE, συζητήσαμε και με την Επίτροπο Μπιενκόφσκα, εμείς ε, ως ε, κοινοβούλιο ε, μπορεί να καθυστερήσουμε τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει ορισμένα δεδομένα να υπάρχουν. Η δημοθεσία RDE θα πρέπει το σε φθινόπωρο του 2017 να εγκριθεί και θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ ουσιαστικά, όχι να πετάμε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Τώρα, για το λογισμικό, για την απάτη, ε, εδώ δεν αναφέρθηκαν ε, πολλά πράγματα. Θα πρέπει να δούμε ε, τις συνειδητές περιπτώσεις απάτης και στις δοκιμές εργαστηρίου και εν χρήση. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση, μία ρύθμιση για τη διαφάνεια η οποία να είναι αποτελεσματική για όλους. Θεωρώ ότι η επικοδομητική συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με τους ε, σκιώδεις ηγητές. Ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο και στη Γερμανία ε, είναι ε, αυτό της, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχαμε καλέσει ε, τον Πρωθυπουργό της Κάτω Σαξονίας που δεν μπόρεσε να έρθει. Τώρα ε, συζητείται ε, η, η, η επίκριση του κυρίου Πύρχε ότι ήδη πριν από το Σεπτέμβριο του 2015 ε, ήταν γνωστή η ε, στάση της Volkswagen στα θέματα αυτά. Δεν είναι σωστό βέβαια να ε, διαπληκτίζονται έτσι. Ο, υπάρχει διάσταση μεταξύ του Πρωθυπουργού κάτω της Αξονίας και του Πύρχια. Ε, εμείς τώρα στις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, δεν είχε προβλεφθεί παράταση, ούτε θα τη ζητήσουμε, αλλά η ερώτησή μου είναι και ίσως μπορούμε να το δούμε ως τους συντονιστές θα πρέπει αυτά στις επί... τις ε, τελευταίες εξελίξεις να τις λάβουμε υπόψη μας στη δουλειά μας και να απευθυνθούμε στους κυρίους Βίλ και Πύρχ ή ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τη γραπτή διαδικασία ενδεχομένως. Ίσως αυτό το κομμάτι των εξελίξεων και της συζήτησης δεν πρέπει να ε, παραγωνιστεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι η κομματική πολιτική σιγά σιγά απομακρύνεται από την Επιτροπή μας, γιατί μπαίνουμε όλο και περισσότερο στις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ο συνηγητής βέβαια δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τη δουλειά μας, για τις τροπολογίες. Ο Γιάννης Κίσκη ανέφερε πολλές τεχνικές λεπτομέρειε της έκθεσης και των τροπολογιών. Τούτου, τούτου δοθέντος, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο, αλλά θα περιοριστώ σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις, σε γενικά σχόλια. Αν δείτε από πού ξεκινήσαμε ε, πριν από ένα χρόνο, ε, ορισμένες πολιτικές ομάδες δεν θέλανε καν την ε, σύσταση της Ερευνητικής Επιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής. Άλλες πολιτικές ομάδες είχαν ήδη καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα πριν καν ξεκινήσουμε την έρευνά μας. Και είδα ότι η παρούσα Επιτροπή ασχολήθηκε με, το, με την ουσία, με το περιεχόμενο και είδα ότι από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά όλοι κινούμαστε, συγκλίνουμε προς έναν κοινό στόχο. Και εγώ ομιλώ σε ένας από τους συντάκτες του σχεδίου έκθεσης, αλλά και ο Γιάννης και ο Παύλο έχουμε καταφέρει να συντάξουμε ένα σχέδιο έκθεσης που οι περισσότεροι από εμάς ε, θα εξέφραζαν την ε, θετική τους γνώμη γι' αυτό. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι βελτίωσης και κάποιες τροπολογίες, πολλές τα έλεγα, πράγματι βελτιώνουν την έκθεση. Ωστόσο, αν και ε, υπάρχουν, το 99% των τροπολογιών δεν αλλάζουν την έκθεση δραστικά. Και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό για εμάς, εμάς που δουλέψαμε 11 μήνες τώρα, ε, για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή έκθεση. Και ο Γιάννης και εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους και οι εισηγητές για τη στενή του συνεργασία για τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί χρειάζεται να συμφωνήσουμε ε, για αυτά. Και αυτά το πετύχαμε πέρσι το Δεκέμβριο. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο στην εξέβρεση των λύσεων, ότι θα βρεθούν λύσεις. Ε, κάποιες δυσκολίες παραμένουν Τελικά θα πρέπει να ψηφίσουμε και θα πρέπει να δούμε το συσχετισμό μη δυνάμεων και ποια πλειοψηφία θα διαμορφωθεί. Όμως με αισιοδοξία ε, περιμένω να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές τις επόμενες εβδομάδες και περιμένω και την ε, ψηφοφορία στα τέλη αυτού του μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, πράγματι ήταν πολύ θετικό το κλίμα και αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω και εγώ να το υπογραμμίσω. Η κυρία Μπόνιφα, σας ευχαριστώ. Και εγώ είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη για αυτή τη συλλογική δουλειά που έγινε και κυρίως επί των αριθμητικών στοιχείων, επί των πραγματικών γεγονότων. Είναι μια δουλειά που έφερε καρπούς και ήταν πολύ σημαντική για να περάσουμε στα συμπεράσματα και στις συστάσεις. Το κείμενο ήταν καλό γιατί η δουλειά της Εξεταστικής Επιτροπής εμείς ήταν πολύ σημαντική. Κατανείμαμε τα καθήκοντα και τις εργασίες πολύ σωστά μεταξύ μας και βλέπουμε ότι είναι σημαντικές και πολλές οι συγκλήσεις. Όλο αυτό είναι ουσιώδες. Ωστόσο, όπως είπε ο Γέντς και ο κύριος Γκεμπράντη, Υπάρχουν θέματα επί των οποίων δεν συμφωνούμε ακόμα και οφείλουμε να το πούμε ανοιχτά, να το παραδεχθούμε και ε, χρειαζόμαστε ε, περισσότερο χρόνο. Ε, οι σκιώδεις εισηγητές συνεδρίασαν χθε και εντόπισαν κάποια τέτοια ζητήματα και ήταν χρήσιμη αυτή η σύσκεψη. Θα χρειαστούν άλλες δύο πιστεύω για να ε, διαλυθούν όλες οι αμφιβολίες. Υπάρχουν ορισμένα σημεία για τα οποία οι σοσιαλδημοκράτες έχουν συγκεκριμένες αμφιβολίες. Θα συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε. Και στην ακρόαση της κυρίας Επιτρόπου αναφερθήκαμε ιδιαίτερο σε ένα από αυτά τα θέματα που είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής. Είναι πολύ απογοητευτική η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το παρόν η οποία λέει ότι παραμένει το θέμα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών όταν όλοι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θέμα αποτελεσματικότητας, ότι τα κράτη-μέλη δεν σέβονται την κείμενη νομοθεσία ε, και αν δεν, τελικά δεν υπάρξει ανεξάρτητη αρχή θα υπάρξουν νέα τέτοια σκάνδαλα τα επόμενα χρόνια. Και στις επόμενες συνεδριάσεις όταν θα συζητήσουμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν υπάρχει σαφής εντολή στο κοινό ερευνητικό ε, κέντρο. Δεν έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή εντολή για να μελετήσει τη μη τήρηση και την, ε, τα συστήματα αναστολής που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές. Ο νόμος εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τη μία χώρα στην άλλη και πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε συστάσεις, όπως το, ε, συστάσεις για αυτό το θέμα, συστάσεις για το καθεστώς των κυρώσεων, για την ανάγκη ε, ενιαίου συστήματος κυρώσεων και απόσυρσης της έγκρισης και της άδειας τελικά, ανάγκη να αποσμειωθεί ο καταναλωτής, και ναι, κυρία Πρόεδρε, άκουσα την κυρία Επίτροπο να λέει ότι σήμερα δεν πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δράσουν, δεν μπορούν να δράσουν ευρωπαϊκά, μπορούν μόνο να παρακινήσουν. Εμείς όμως έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και νομίζω ότι όλοι οι παρόντες το συμμερίζονται αυτό. Ότι εμείς ε, ε, ε, είμαστε εξαιρετικά σε γρηγόρση για θέματα προστασίας του κατάλωτη. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάληψης ευθυνών όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να υπάρξει παράγοντας που θα συμβάλλει στη συμμόρφωση το συντομότερο δυνατό. Οι εξεταστικές επιτροπές μπορεί να διευκολύνουν το έργο τους. Δεν έχει ακολουθηθεί το σωστό χρόνο διάγραμμα στις εργασίες της Ερευνητικής και Εξεταστικής Επιτροπής και θα ήθελα την πρότασή μας να τη όλοι, έτσι ώστε η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και η ψήφιση ε, στην Ολομέλεια ε, του κειμένου για τα σωματίδια να λάβει χώρα την ίδια στιγμή. Δηλαδή να υπάρξει συγχρονισμός μεταξύ των δύο αυτών ε, πρωτοβουλειών ε, της διαδικασίας με την οποία θα εγκριθούν στις αρμόδιες επιτροπές και στο, στην Ολομέλεια. Όλα αυτά πιστεύω ότι τα συμμερίζονται οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και το λέμε από την αρχή της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Το διακύβευμα είναι μεγάλο και η ευθύνη της Επιτροπής μας εξίσου μεγάλη. Δεν είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε μόνο, αλλά για να κάνουμε συστάσεις και πιστεύω ακραδάντως ότι όλοι συμφωνούν ότι καλώς υιοθετούμε μια συνολική προσέγγιση του κλάδου ε, λαμβάνουμε υπόψη μας τις θέσεις απασχόλησης και την έρευνα και την τεχνολογία Λαμβάνουμε υπόψη μας την υγεία του Ευρωπαίου καταναλωτή, την ανάγκη προστασίας της υγείας αυτού και του περιβάλλοντος, η συνολική λοιπόν ολική προσέγγιση η οποία πρέπει να υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα πρέπει οι προτάσεις μας να υποβάλλονται σε άλλο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των κρατών μελών. Μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, η ευρωπαϊκή βαθμίδα είναι αυτή που θα κομίσει την αναγκαία και επιπρόσθετη ε, προστασία. Είναι ε, εξόχως πολιτικό ζήτημα να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τους καταναλωτές σε όλες τις διαστάσεις της ζωής τους, ε, στην καθημερινότητά τους και υπ' αυτή την έννοια πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να συμβάλλουμε ε, για την υποβολή συμβαστικών τροπολογιών, που, τις οποίες θα προσυπογράψουμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Χιάνκελ, ο σκιώδης για το ECR, δεν είναι παρόν. Θα ήθελα να πάρω το λόγο τώρα εγώ στη θέση του, να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την εξαιρετική εργασία που έχουν κάνει και προσβλέπω και εγώ στις μελλοντικές συζητήσεις που θα διεξαχθούν. Τώρα το σχέδιο συμπερασμάτων μας βρίσκει σύμφωνους, στέλνει ένα πολύ χειρό πολιτικό μήνυμα και καλύπτουν όλους τους τομείς τα συμπεράσματα αυτά. Έχω υποβάλει βέβαια κάποιες τροπολογίες μαζί με την Τζούλη Gerling θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία λοιπόν σημεία, αν μου το επιτρέπετε, και τα όσα θα πω συνδέονται με τα ζητήματα τα οποία θέσαμε ως ερωτήματα και παρατηρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα οποία δυστυχώς απάντηση δεν πήραμε. Στην τροπολογία 28 ζητούμε καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση για τους καταναλωτές. Επί μακρόν το συζητήσαμε αυτό. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση προς τους καταναλωτές θα πρέπει να βελτιωθεί και να διευρυνθεί. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων, όσον αφορά τα μικροσωματίδια και όσον αφορά το μονοξίδιο του αζότου και θα πρέπει να διεξαχθεί και ένας διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κλάδου και των κρατών μελών γιατί όπως καταλαβαίνετε το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι ένα ζήτημα κοινό που αφορά τους πάντες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και ο κλάδος θα πρέπει να λάβει το ρόλο του στον τομέα της δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, το όλο το περιεχόμενο πλέον των απαιτήσεων που προβάλλουμε προς τα κράτη-μέλη και προς τον κλάδο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διαγραμματίσουν τον ρόλο τους προκειμένου να προωθηθεί περισσότερο η κυκλοφορία των οικολογικών αυτοκινήτων. Έχουμε και μία ακόμα τροπολογία που έχουμε καταθέσει και που συνδέεται επίσης και με την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ όσον αφορά το σύστημα έγκρισης τύπου είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία υπηρεσία παρακολούθησης ευρωπαϊκή όσον αφορά τα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτού υπάρχει η κοινή συνένεση, όπως έχετε δει στην Επιτροπή μας, και το θέλουμε αυτό γιατί θέλουμε μια πιο ανεξάρτητη αρχή επιτήρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημιουργίας, της θέσπισης ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού επιτήρησης αγοράς. Το είπανε και αυτό και οι δύο συνεισηγητές οι οποίοι ε, απευθυνόμενοι στην εφημερίδα EU Observer είπαν ότι δεν ήταν απόλυτα πεπισμένοι για την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας ε, ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής. Και ότι αν δημιουργείται τέλο πάντων μια τέτοια αρχή θα ήταν σαν να λέμε ότι δεν εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι αν μάθαμε κάτι από την εξαστική μας Επιτροπή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έπραξε σωστά, ότι υπέπεσε σε πάρα πολλά λάθη, ότι σε άλλε περιπτώσει δεν ανέλαβε επαρκή δράση. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο εμεί θεωρούμε ότι είναι απόλυτα θεμητό το να πετούμε να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή και ελπίζουμε ότι οι τροπολογίε μα αυτέ θα ενταχθούν στο τελικό κείμενο. Είμαι εξουσιοδοτημένη να μιλήσω για τον σκιώδη μας και την ομάδα και να πω τη θέση μας. Δεν ξέρω αν είμαστε στην αρχή ή στο τέλος της Επιτροπής. Μου φαίνεται ότι είμαστε στη μέση. Διαπιστώνουμε ότι έχουν παραμείνει πολλά άλυτα θέματα. Και δεν είναι αλήθεια ότι δεν ήξερε κανείς τίποτε. Πολλοί το ήξεραν εδώ και καιρό, είχε ενημερώσει και η περιβαλλοντική υπηρεσία στη Γερμανία είχε έρθει σε επαφή με τη γερμανική κυβέρνηση για να ενημερώσει για τα θέματα που αφορούσαν το σκάνδαλο των εκπομπών και υπήρχαν και πληροφορίες που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε δεν μπορεί κανείς εύκολα να ισχυριστεί ότι κανείς δεν ήξερε τίποτε. Ε, δεν είμαι βέβαιη αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με το ΕΛΚ σε όλα τα θέματα. Ε, σε ορισμένα σοβαρά θέματα διαφοροποιούμε θα εμείς και θέλουμε περισσότερη συνέπεια. Περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι μόνο να ανακαλύπτουμε τις απάτες και να ανακτούμε τη χαμένη εμπιστοσύνη, παρόλο που αυτό είναι σημαντικότατο βέβαια, πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων, την περιβολαντική προστασία, τους στόχους που θέσαμε εμείς οι ίδιοι και για την τήρηση του ενωσιακού δικαίου. Και ε, αυτά σημαίνουν πολλά. Υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία συμφωνούμε στην έκθεση, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για την Κομισιόν. Η Κομισιόν και και τα κράτη-μέλη απέτυχαν. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, αφού διαπίστωσαν τις ε, ε, διαφορές το 2013 ενημερώθηκαν για την, τις διατάξεις αναστολής που χρησιμοποιούνται και δεν αντέδρασαν. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Η Κομισιόν δεν είπε ξεκάθαρα τι θα μπορούσε να είχε κάνει με βάση το ρόλο που έχει και δεν άσκησε τον εποπτικό της ρόλο όπως έπρεπε δεν είναι μόνο συντονιστής η Κομισιόν ε, μεταξύ των ε, εμπλεκομένων, των διαδίκων, αλλά είναι και θεματοφύλακας των συνθήκων και θα πρέπει να φροντίζει για την εφαρμογή των οδηγιών και της νομοθεσίας εν γέννη. Και μου φαίνεται ότι αυτό δεν το έκανε. Διαπίστωση. Ξεκάθαρη. Ε, επέριψε την ευθύνη στα κράτη-μέλη, τα οποία είναι συνυπεύθυνα σίγουρα, ε, σε ό,τι αφορά το, την υπόθεση αυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, πρέπει να γίνεται και αυτοκριτική, πολύ σημαντικό. Ο μεγάλος χαμένος σε όλη αυτή την υπόθεση και πρέπει να το λέει αυτό καθαρά η έκθεση είναι οι καταναλωτές οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε αυτή την διαπλοκή μεταξύ πολιτικής και οικονομίας ε, και η Ευρώπη υπολείπεται σε θέματα αποζημιώσεων όπως είπαμε. Και δεν έχει σημασία αν κάποιος πρωθυπουργός από την, ε, τους σοσιαλδημοκράτες ε, εμπλέκεται ή κάποιος ε, χριστιανδημοκράτης που θα πάει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Λίγα, πολύ λίγα πράγματα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Αυτά ήθελα να αποτυπωθούν. Αυτό που είναι σημαντικό και με τις τροπολογίες μας το επιχειρήσαμε είναι το πρώτο, να υπάρχουν ε, σαφείς κανόνες για τη δουλειά των lobbyists. Ε, είναι ένα γενικότερο θέμα αυτό που αφορά και άλλες επιτροπές, αφορά όλες τις δραστηριότητές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λέμε εδώ ότι θα πρέπει να ε, ισχύουν οι κανόνες ε, και θα πρέπει να αναφερθεί αυτό και στη συγκεκριμένη έκθεση. Εμείς λέμε σαφώς ότι για τις επόμενες εξεταστικές και το έργο τους θα πρέπει να έχουμε σαφείς διατάξεις, στιβαρές, ούτως ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να ανταποκρίνεται στην αποστολή του, δηλαδή να κάνει έρευνα. Η σύσταση της ε, ΕΜΙΣ έγινε σε μια εποχή όπου ήδη είχε αρχίσει να ε, γίνεται η νομοθετική εργασία. Ε, εμάς μας ενόχλησε πάρα πολύ και πρέπει να το πω αυτό ότι η συνεργασία ε, πολλές φορές ε, ήταν καταστροφική ε, ε, με καθυστερήσεις, με, με απουσίες και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο βέβαια παρατηρείται αυτό πρέπει να πω γιατί πολλές φορές οι εμπειρογνώμονες δεν ε, ε, συμμετέχουν και στην, ε, στην, στις εξεταστικές επιτροπές για τις, τα σκάνδαλα με τις εκπομπές. Τόσο πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί η Επιτροπή μας. Η διαφάνεια επίση είναι σημαντική, η ταχύτητα ε, στην υποβολή των εγγράφων που ζητούνται και ε, πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας και το ε, ζητούμε αυτό μετεπιτάσεως είναι να μπορούν και οι βοηθοί μας να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα ούτως ώστε να προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τον κύριο Γκεμπράντη και τον κύριο Κίζεσεκ. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Οι ευθύνες σας είναι πολύ μεγάλες, γιατί εσείς είστε οι εισηγητές. Η έκθεσή σας θα στείλει μήνυμα προς τα έξω και άρα προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό το Dieselgate δεν συντάραξε μόνο τα κράτη-μέλη και την ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Συντάραξε και τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε εμάς, σε αυτό που κάνουμε εμείς ως πολιτικοί ηθήνοντες, ως και βλέποντας το χρονοδιάγραμμα εκφράζω τη λύπη μου διότι η έκθεση για το Type Approval της εγκρίσης τύπου ε, ψηφίζεται στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, ενώ τα δικά μας συμπεράσματα δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Υπάρχει πρόβλημα επί της ουσίας, αν θέλετε, από πλευράς χρονοδιαγράμματος και νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, αγαπητοί εισηγητές, θα ήθελα να εξετάσετε σε βάθος την εξαιρετική δουλειά της Επιτροπής ΕΜΒΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτές οι δύο επιτροπές ανοίγουν δρόμους, δίνουν κατευθυντηρίες γραμμές στη δουλειά μας. Πολλοί από εσάς μιλήσατε για την περιβόητη ανεξάρτητη αρχή υπηρεσία ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει το ενδεχόμενο της σύστασης. Μια πιο μετριασμένη διατύπωση. Σας συγχαίρω αγαπητοί εισηγητές γιατί αναλαμβάνετε την ευθύνη και λέτε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνες, όμως όπως είπε και η Επίτροπος προλίγου, Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν αντλήσει τα διδάγματα που τους αναλογούν μετά από αυτό το σκάνδαλο. Θα πρέπει η έκθεσή σας να τονίσει ακόμα περισσότερο τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντλήσει διδάγματα από αυτό το σκάνδαλο. Έχετε δίκιο κύριε Σιγητά όταν το λέτε. Και γι' αυτό εμείς υποβάλλουμε την τροπολογία υπαριθμών 47, η οποία λέει ότι αν δεν έχει γίνει σωστή χρήση των πληροφοριών που διαχειρίζεται το κοινό ερευνητικό κέντρο μεταξύ 2000, 2009 και 2010 και θα έπρεπε να είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο παρουσίας ε, παράτυπου και παραπλανητικού λογισμικού. Ε, λέει περίπου αυτά και παραθέτω ε, το απόσπασμα. Επομένως, κύριοι συγητές, θεωρώ ότι η έκθεσή σας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορεί να δείξει ότι πρέπει να υπάρχει ένα πριν και ένα μετά το σκάνδαλο Ντίζελ και να είναι ξεκάθαρα ε, ε, διαχωρισμένα αυτά τα δύο. Ε, συμφωνούμε όλοι στην Εξεταστική μας Επιτροπή να μην ξαναυπάρξει Dieselgate στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να, υπά... να συμπεριληφθούν και θα προσέξω ιδιαίτερο στη συνέχεια που θα δοθεί και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ. Η κυρία λόγο. σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο εισηγητές μας οι οποίοι μολονότι υπήρχαν διάφορες αμφιβολίες και ως προς την αποτελεσματικότητα της Εξεταστικής μας Επιτροπής τελικά, τελικά πρέπει να πω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και τα δύο κείμενα και οι δύο εκθέσεις περιλαμβάνουν πάρα πολλά από τα κρίσιμα αυτά σημεία, τα οποία εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των ακράσεων που είχαμε τους δύο τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, το ζήτημα της ενιαίας αυτής ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Αρχής. Να πω και εγώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάχθηκε αυτή υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου ανεξάρτητου οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να ασχολείται με την επιτήρηση της αγοράς. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν προκειμένου να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και εμείς. Όντω, ε, η Επιτροπή ΙΜΚΟ και κάποιε άλλε επιτροπέ που εκνοδομοτούν στο Κοινοβούλιο έχουν πολύ πιο ήπια στάση. Α μην επηρεαστούμε από αυτέ. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει ως εξεταστική επιτροπή να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί. Ούτω ή άλλω η έκθεσή μα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Κάνει συστάσει, καταλήγει σε συμπεράσματα. Ένα ακόμα σημείο. Όσον αφορά του συντελεστέ συμμόρφωση, Ασχοληθήκαμε ως ασκιώδη ηγητές και με το ζήτημα αυτό. Στις πρώτες δοκιμές που είχαμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, όπως φάνηκε άλλωστε από τις πρώτες δοκιμές, έναν συντελεστή συμμόρφωσης ο οποίος να μπορεί να πλησιάζει τη μονάδα χωρίς να προβλέπονται άλλες διατυπώσεις ή άλλο περιθώριο ευελιξίας όπως είχαμε στο παρελθόν ο στελεστής συμμόρφωσης θα πρέπει να βαίνει προς τη μονάδα και να μην δεχόμαστε κάποια άλλα, διαβάθμιση, κάποια άλλα πέρα από αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σωρίνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και να σας υπενθυμίσω λίγο το πνεύμα της κοινή εργασίας που χαρακτήρισε την εξεταστική μας αυτή επιτροπή και που μας επιτρέπει τώρα να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που μπορεί τελικά να μην έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τα πάντα, αλλά έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Προφανώς θα πρέπει να συνεχιστεί η εργασία μας μέχρι την τελική έγκριση των δύο αυτών εκθέσεων. Καταφέραμε εμείς να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για την ίδια την αυτοκινητοβιομηχανία, θα έλεγα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ε, πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο την εργασία αυτή στο μέλλον. Είναι σαφές ότι δεν υπήρξε απαραίτητη πολιτική βούληση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να τηρήσει εντελώς την εντολή της δηλαδή και να κατακρίνει, να αποδοκιμάσει και να αποτρέψει τις ε, απατηλές πρακτικές ε, των ε, κρατών μελών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές, τα πραγματικά στατιστικά δεδομένα όσον αφορά το επιτρεπόμενο επίπεδο μόλυνσης του περιβάλλοντος και ποιες είναι οι μετρήσεις τελικά που γίνανε για να αποφευθεί αυτό σε εργαστηριακό επίπεδο και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εμείς να επικρίνουμε και να αποδοκιμάσουμε την όλη αυτή νοοτροπία που είχαν τα κράτη-μέλη και η αυτοκινητοβιομηχανία. Μία νοοτροπία μη ανάληψη ευθυνών, ανευθυνότος θα έλεγα, και αυτό το είδαμε πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει και να ενισχύσουμε την εντολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών και να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή για την επιτήρηση της αγοράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις παραλυθούσες αυτές πρακτικές, οι οποίες λειτουργούν κατά των Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν καν την επαρκή αποζημίωση, όπως είδαμε. Επικεντρωθήκαμε στα πλαίσια της εργασίας μας σε όλα αυτά τα σημεία και αυτή είναι η δική μου προσωπική σκοπιά τώρα, αν θέλετε. Επ' αυτού όμως νομίζω ότι συμφωνήσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε εν πάση περιπτώσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Να επανέλθουμε στους εισηγητές. Ο κύριος Γκεμπράντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω λεπτομερώς σε όλες τις παρεμβάσεις γιατί από ό,τι κατάλαβα μου εξέφρασαν οι ομιλητές τη στήριξή τους ε, στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο του συνεισηγητή και τους ευχαριστώ πολύ. Ε, επειδή τέθηκε συγκεκριμένο ερώτημα για την υπηρεσία αυτή, θα ήθελα να απαντήσω. Δεν είναι ότι είμαι κατά. Δεν είμαι κατά επί της αρχής της ε, αυτόνομης αυτής υπηρεσίας και γι' αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στήριξα την άποψη των συναδέλφων και πριν μάθω περισσότερα, στήριζα την ε, πρόταση σύστασης αυτόνομης υπηρεσίας. Ωστόσο, δεν, ε, έχω κάποιες εντηρήσεις, θεωρώ, ότι δεν θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να συσταθεί ε, μέσα στα απόνερα του Dieselgate. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε, την, έχουμε εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, είναι ισχυρή, είναι δυνατή και ελέγχει την εφαρμογή ε, των νόμων μέσα στα κράτη-μέλη. Και αυτό υπάρχει στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρος. Από τη στιγμή λοιπόν που λέμε ότι η δεν εμπιστευόμαστε επιτέλους και πια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των εκπομπών των σωματιδίων, των ρήπων και ούτω καθεξής και θέλουμε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αυτόνομο φορέα άλλο, τότε υπονομεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα την Ευρωπαϊκή Ένωση εσύ θέμελα και στο σύνολό τους. Πρέπει λοιπόν να λέμε ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύουμε για την ίδια. Θα, το λογικό συμπέρασμα δηλαδή θα πρέπει να είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεξαρτησία της και όχι απαραίτητα να δημιουργηθεί κάτι το ανεξάρτητο γιατί είναι σαν να λέμε ότι η Επιτροπή δεν έχει ε, ανεξαρτησία ή δύναμη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να ενισχύσει το ρόλο της ε, και για τα σωματίδια και για την, ε, ε το, το, την τήρηση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Ο... Όντως ε, η εικόνα των κρατών μελών είναι πολύ δυσάρεστη και της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης. Αλλά μας υπόθηκε ότι δεν ήξερε τι ακριβώς να κάνει και έτσι είναι σαν να δώσαμε επιταγή λευκό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν νομίζω ότι μια αυτόνομη υπηρεσία θα λύσει το θέμα. Πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες πρωτοβουλίες. Είναι θεσμικό όργανο, κοινό για όλους μας. Επανειλημμένος. Έχουμε πει ότι ήδη έχουμε μια τέτοια υπηρεσία για όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και για τις οδικές μεταφορές, αλλά όχι ως αποτέλεσμα του Dieselgate. Η κυρία Μπονίφα, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Γκεμπράντη. Θέλω όμως να σας καθησυχάσω. Όταν προτείνουμε τη σύσταση μιας υπηρεσίας τέτοιες, δεν αμφισβητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε μεριμνούμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να δράσει. Αντιθέτως, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα. Και αυτό είχε πει και ο συνάδελφος και με, πάνω σε αυτή τη βάση είχα προτείνει την ιδέα στην πολιτική μου ομάδα. Έχουμε την ΕΡΑ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η οποία υπάρχει όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ασχοληθεί, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το, ο εκτελεστικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η υπηρεσία ενδιαφέρεται για τον έλεγχο, τη διαιτησία των σιδηροδρομικών μεταφορών και ενδεχομένω την επιβολή κυρώσεων μετά από συνένεση και συνέργεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση μη τήρηση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά δεν είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό, ούτε αμφισβητείται ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσατε για την υπηρεσία οδικών μεταφορών. Σε ένα ψήφισμα πρόσφατο, το ψήφισμα κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, ε, ψηφίσαμε την επιθυμία μας να υπάρξει μια υπηρεσία αυτόνομη για τις χερσαίες μεταφορές. Και από τη στιγμή που έχουμε ήδη υπηρεσία για τις υδροδρομικές μεταφορές, μπορεί κανείς να φανταστεί ε, οι αποστολές τους να ε, πηγαίνουν χέρι-χέρι των δύο αυτών υπηρεσιών. Δεν το λέμε και δεν το προτείνουμε γιατί δεν εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά γιατί θέλουμε καλύτερα να διευκρινιστούν οι ρόλοι και τα καθήκοντα και σιγά σιγά να βρεθεί συνέργεια και συμφωνία μεταξύ των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ρωτήσαμε ε, στη δική μας Εξεταστική Επιτροπή μας είπαν τα περισσότερα εξ αυτών ότι είναι υπέρ αυτού του ενδεχομένου. Να καθισχάσουμε δηλαδή την Επίτροπο ότι δεν αφιζητούμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα διασφαλίζει ότι η νομοθεσία τηρείται παντού στην Ευρώπη. Θέλουμε να βεβαιωθούμε όμως ότι σωστά ερμηνεύεται ο νόμος παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Δεν έχει κλείσει αυτή η συζήτηση ακόμα θα έχετε και άλλες συζητήσεις στις συναντήσεις και συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Γκίζεκ, ευχαριστώ. Είναι ειδική αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Έχουμε συνεισηγητές που συνεργάστηκαν πολύ καλά. Άλλωστε συνόψησε ο συνάδελφος τόσο καλά τα θέματα που δεν ε, έχω πολλά να πω. Ένα λεπτό μόνο. Και εγώ πριν από ένα χρόνο δεν θα φανταζόμουν ότι θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Ε, προσεγγίσαμε ένα τον άλλον, συνεργαστήκαμε καλά και τώρα ε, ε, ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εις ό,τι αφορά τον ενίο ευρωπαϊκό οργανισμό, ε, θα έπρεπε να το δούμε καλύτερα. Αν δούμε ε, ότι θα συζητηθεί το θέμα και θα διαφοροποιηθεί η άποψη των επιτροπών, ε, όταν η Κομισιόν και το Συμβούλιο δουν τη δουλειά μας, θα πούν ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχουν 97 διαφορετικές γνώμες για το θέμα του νέου οργανισμού. Δεν είναι καλό αυτό και δεν μας εξυπηρετεί. Πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικά. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, πρέπει να έχουμε τεκμηριωμένες απόψεις. Και στο τέλος, και όπως είπε και η κυρία Ντελή, όταν ε, εγκρίνουμε τις συστάσεις και ψηφίσει και η ΙΜΚΟ για τα θέματα αυτά, ε, δεν θα, ε, αν μείνουμε εδώ που είμαστε, δεν θα έχουμε συνέπεια πρέπει δυνατόν να μιλήσουμε με μία φωνή. Στο θέμα του οργανισμού, δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία άποψη. Ω ένα βαθμό συμμερίζομαι και το επιχείρημα του κυρίου Γκερμπράντι ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ε, έχουμε δυσπιστία προς την Κομισιόν. Ε, δεν είναι πάντα ε, λύση ο ένας νέος οργανισμός. Μέχρι να γίνει το να, να, συσταθεί, να ε, υπάρξει, να προσληφθεί το προσωπικό, ε, να ληφθούν οι αποφάσεις, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Πρέπει να ενισχύσουμε την Κομισιόν λοιπόν και όχι να μεταθέσουμε τις ευθύνες σε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό. Προσοχή λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσει με μία φωνή. Πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Έχουμε 6-7 μέρες στη διάθεσή μας μέχρι τις 28. Ε, το ΕΛΚ θα συνεργαστεί επικοδομητικά ε, και ε, ήδη έχουμε και πολύ καλή, είχαμε και ευχαριστώ γι' αυτό πολύ επικοδομητική συνεργασία από όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά πρέπει να πω. Ε, οι συγητές και οι σκιώδεις έχουν ε, ακόμα λίγη δουλειά να κάνουν. Στις 28 Φεβρουαρίου πρέπει να ψηφίσουμε. Ίσως θα πρέπει να ε, δούμε και τα, τις τελευταίες γερμανικές εξελίξεις, Μπορείτε να ενημερώσετε με email τη γραμματεία σχετικά. Θέλετε να πείτε κάτι μετά. Θα ήθελα να μην παραταθεί η ε, διάρκεια της Επιτροπής, η λειτουργία της Επιτροπής, να προχωρήσουμε, να ψηφίσουμε και να το τελειώσουμε. Και μπορούμε να πάρουμε κάποιες προσθήκες γραπτός και μετά θα ενημερωθώ και από τους ε, συντονιστές. Όχι, όχι, όχι, δεν ήθελα να ζητήσω παράταση της, της εντολής. Στα πλαίσια του 12 μήνου ε, έπρεπε να καλύψουμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τη Γερμανία. Θα στείλω mail και ε, ή θα ζητήσω έκτακτη συνεδρίαση ή θα ακολουθήσουμε την γραπτή διαδικασία. Ο κύριος Γκερμπράντι. Διαφορετικό είναι το δικό μου το αίτημα, κυρία Πρόεδρε. Χθε από τη γραμματεία μας ενημερωθήκαμε ότι ε, ως Επιτροπή λάβαμε περισσότερα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια περαιτέρω έγγραφα τα οποία είναι εμπιστευτικά και βρίσκονται στην αίθουσα αυτή, την ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης. Πρόκειται για έγγραφα από συνεδριάσεις ε, του Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του 2016. Μου κάνει εντύπωση ότι τα πρακτικά από τον Απρίλιο του 2016 τα λαμβάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο τώρα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο λαμβάνουμε λοιπόν τα πρακτικά αυτά μόνο τώρα, μόνο ότι εμεί τα είχαμε ζητήσει μετά τη συνεδρίαση τη 12η Μαου. Την επόμενη εβδομάδα πάμε στο Στρασβούργο, την επόμενη εβδομάδα ψηφίζουμε, όπω είπατε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να συμβολευτούμε τα εμπιστευτικά αυτά έγγραφα και με όλου του άλλου περιορισμού που έχουμε και με του περιορισμού που υπάρχουν ω προ το ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την αίθουσα ανάγνωση... τα πράγματα δυσχεραίνονται ακόμα περισσότερο. Ένα ακόμα αίτημα. Δεν έχουμε λάβει ακόμα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία τα έχουμε ζητήσει του τελευταιου 12 12-13 μήνε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα συνολικό κατάλογο από τη γραμματεία μα Ποια έγγραφα περιμένουμε ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εσεί ω πρόεδρο μπορείτε να ασκήσετε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα αυτά. Όχι τον επόμενο μήνα όμω γιατί ψηφίζουμε τέλη Φεβρουαρίου. Και αφού ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τα τέλη Φεβρουαρίου, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε πλέον να τροποποιήσουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί δεν μπορούμε να υποβάλουμε, όπως ξέρετε, περισσότερες τροπολογίες στην Ολομέλεια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να λάβουμε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού ψηφίσουμε εδώ πέρα και ή δυνατόν όχι μία ώρα πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προωθήσω τα αιτήματά σας αυτά και θα σκίσω πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία ακόμα φορά. Ο κύριος Νέιμαρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο, στην αίθουσα. Μπορείτε ενδεχομένω να μας πείτε εσείς για ποιο λόγο έχουμε τόσο σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την τεκμηρίωση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Σας διαβεβαιώ ότι κάνω κάθε, κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να προσκομίσουμε τα έγγραφα αυτά τα οποία ζητήσετε το συντομότερο δυνατό. Όπως ξέρετε, λειτουργούμε στα πλαίσια ενός ε, δύσκολου περιβάλλοντος κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με έγγραφα στα οποία μπλέκονται και τρίτα μέρη. Και αυτό συμβαίνει ιδίω με τα έγγραφα αυτά της TCMV, της Τεχνικής Επιτροπής για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα, που πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με άλλους εμπλεκομένους. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση αυτή για μας. Ε, χρειάζεται αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουμε κάποια έγγραφα τα οποία δεν συνηθίζουμε συνήθως να ζητάμε, να προσχομίζουμε. Ενδεχομένως αυτό να απαντά εν μέρη στο για ποιο λόγο δεν έχουν φτάσει, μόλις τώρα φτάνουν κάποια πρακτικά από παλαιότερες συνεδριάσεις της ε, TCMV. Δεν εξαρτάται άμεσα από εμά. Επίσης δεν γνωρίζαμε ότι θέλατε το σύνολο των πρακτικών. Αυτή τη στιγμή λάβαμε το αίτημα αυτό, αρχίσαμε να προωθούμε όλα τα έγγραφα. Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εκκρεμούν αυτή τη στιγμή κάποια αιτήματα για έγγραφα τα οποία ενδεχομένω να μην έχουμε ακόμα προσκομίσει ή για τα οποία δεν έχουμε δώσει ακόμα κάποια πρώτη απάντηση τουλάχιστον. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν εκκρεμούν ακόμα κάποια αιτήματα τη Επιτροπή σα, το εξετάσουμε τότε περισσότερο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ήδη λοιπόν αυτή την εβδομάδα μπορούμε να προωθήσουμε και προς εσάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τους νηστές όλα αυτά τα αιτήματα τεκμηρίωσης τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Και σας παρακαλώ πολύ ας εισακουστεί το αίτημα του κυρίου Γκερμπράντη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό για μας. Έχουμε κάνει εκτενέστατες συζητήσεις για την ανάγκη εξέτασης των εγγράφων αυτών και από τη δική μας την Επιτροπή. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ επιτρέψτε μας να ολοκληρώσουμε την εξέταση των εγγράφων αυτών πριν την ψηφοφορία μας εδώ στην Εξαστική Επιτροπή. Του των λεχθέντων, ήδη τη Δευτέρα στο Στρασβούργο, ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα προς εξέταση στο Στρασβούργο, προβλέπεται μία συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΑΦΚΟ σε σχέση με την, τα δύο αυτά έγγραφα τα δικά μας. Επομένως, μπορείτε να συμμετάσχετε και στην συνεδρίαση που θα γίνει στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε στα πλαίσια της συζήτησης αυτής που θα γίνει στο Στρασβούργο να δούμε ποιες είναι οι δικές μας εξουσίες, οι αρμοδιότητες που έχουμε, που θα έπρεπε να έχουμε ως Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορούμε, αν μη τι άλλο, με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει εμείς, να θέσουμε κάπως τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για τις εργασίες μελλοντικών εξεταστικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη συνεργασία σας. Ξέρω ότι έχουμε ακόμα δουλειά ως συνεισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για να ολοκληρώσουμε την όλη εργασία μας. Θα σας δω πάλι όλους σαφώς τη συνεδρίαση που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, όπου θα ψηφίσουμε και τα δύο αυτά έγγραφα. Σας ευχαριστώ πολύ.